Benvenuti Καλώς ήρθατε όλοι. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν προσεφέρθη να μας ενημερώσει πριν από την επίσημη διαβίβαση προς το Κοινοβούλιο την, σχετικά με την νέο σχέδιο πρότασης της Κομισιόν για την παρουσία ιχνών γενετικά τροπομένων οργανισμών στα τρόφιμα. Ο κανονισμό θα υιοθετηθεί τι επόμενε μέρε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα εξετάσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης με τα ελέγχου. Μια, μια διαδικασία επιτροπολογίας στην οποία συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Προτείνω λοιπόν να προσθέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και να το εξετάσουμε πριν να ξεκινήσουμε το σεμινάριο για την κοινή γεωργική πολιτική. Αν συμφωνείτε, να εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη με αυτήν την αλλαγή. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ. Ανακοινώσεις. Η σημερινή συνεδρίαση θα αναμεταδίδεται στο web stream, σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη, αντίσταση στα αντιβιωτικά, υιοθέτηση της προφορικής ερώτησης. Οι συντονιστές αποφάσισαν να θέσουν μια προφορική ερώτηση για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Η προφορική ερώτηση έχει μεραστεί στα μέλη της Επιτροπής. Οι συντονιστές επίσης αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να συνοδεύει την προφορική ερώτηση ένα σχέδιο ψηφίσματος που θα προέρχεται από την Επιτροπή μας. Το θέμα λοιπόν αυτό θα περάσει από την Ολομάλεια τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι υιοθετείται η προφορική ερώτηση. Σημείο 4. Τροποποίηση του κανονισμού ΕΕ 1234 του 2007 του Συμβουλίου που αφορά τις ε, συμβατικές σχέσεις στο τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο εισηγητής είναι ο James Nicholson. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως θα θυμάστε, μετά από την κρίση στον τομέα του γάλακτος το 2009 η Κομισιόν πρότεινε μια σειρά νομοθετικών μέτρων που στόχο έχει να σταθεροποιήσει την αγορά εξισορροπώντας την προσφορά και τη ζήτηση χάρη σε μια ενίσχυση των συμβάσεων ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μεταποιητές να σταθεροποιήσει τα εισοδήματα των, παραγωγών ενισχύοντας ε, τα συλλογικά τους διαπραγματευτικά ε, ε, τη δική τους ε, θέση στον τομέα της, ε, του γάλακτος και τέλος να ενισχύσει τη διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αν και αυτές οι προτάσεις ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση, παραμένουν πολλά ακόμα προς αποσαφήνιση. Γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον James που μόλις έφτασε. για να ξεκινήσουμε ένα πρώτο γύρο ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το θέμα. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν και μετά από την παρέμβαση του James Νίκολσον θα ακολουθήσει η συζήτηση. Γι' αυτό όποιος θέλει να πάρει το λόγο να το πει στη γραμματεία. James, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι γενικά οι προτάσεις αυτές έγιναν θετικά, έτυχαν θετική υποδοχή ε, στους ε, οικονομικούς κλάδους. Ε, ε, συνάσαν διάφορους ενδιαφερόμενους από διάφορους τομείς της βιομηχανίας αυτής του οικονομικού κλάδου γενικά και εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις και ορισμένες μάλιστα από τις μόνιμες αντιπροσωπείες εδώ στις Βρυξέλλες. Όπως είπα, οι αντιδράσεις γενικά είναι θετικές, αλλά εξετάζοντας κανένα στις λεπτομέρειες της πρότασης, μπορούν νομίζω να διευκρινιστούν κάποια σημεία και να βελτιωθούν κάποια άλλα. Η πρόταση αυτή θα βοηθήσει την, ε, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ο κλάδος μετά το 2015. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν στον γαλακτοκομικό τομέα μετά από αυτή την προθεσμία. Στι γενικέ ήθελα να παρουσιάσω μέσα από τι σκέψει μου, γιατί προσπαθώ να είμαι ανοιχτό ω συγητή και να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω όμω εγώ ίσω τέσσερι πτυχέ. Καταρχήν τι συμβάσει. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο οι παραγωγοί χρειάζονται τις συμβάσει αυτές. Ήταν να υπάρχουν αντιδράσεις ε, από πολλέ οργανώσει παραγωγών. Αυτή τη στιγμή η πρόταση όμως ε, είναι θελοντική σε εκούσια σε επίπεδο κράτου μέλου. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δείξουν κάποια ευελιξία όπως χρειάζονται. Πολλά αυτά θα με ενδιαφέρε να μου πείτε ποια από τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν αυτή την επιλογή. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεύτερα, όροι και προποθέσει των συμβάσεων θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ο όγκο, αποκλειστικότητα παραγωγή, τιμή, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει το κείμενο να το εγκαταπτύσσει σωστά. Η σκέψη μου θα ήταν να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε κατά δυνατόν ευελιξία όσο περισσότερο μπορούμε να επιτύχουμε. Μία επιλογή θα ήταν να επιστρέψουμε στην αρχική εκδοχή του κειμένου, όπου κάποιος θα, ήθελε να, θα μπορούσε να ζητήσει μία σύμβαση αν το επιθυμούσε. Ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτική η σύμβαση αυτή στο εν λόγω κράτος μέλος. Αυτό είναι ένα θέμα που θα εξετάσω ενδελεχώς. Δηλαδή για τη συμβάση θα πρέπει γενικά να ξέρουμε πού θα μπορούν και θα πρέπει να εφαρμοστούν και ποιοι θα είναι οι όροι τους. Κατόπιν οργανώσει των παραγωγών. και τις δυνατότητες που έχουν για διαπραγματευτική ισχύ μαζί με την ιδέα της αγωγής των ε, συμβάσεων. Αυτό είναι νομίζω το επίκεντρο της πρότασης. Ε, Καταλαβαίνω πού προέρχεται αυτό και αν εξετάσουμε τους κύριου στόχους της πρότασης θα δούμε ότι είναι ακριβώς να ενδυναμώσουν την ισχύ των γαλακτοπαραγωγών για να μπορέσουν να πετύχουν και να βελτιώσουν αυτοί που έχουν διαπραγματευτικού τους ε, θέση. Και εδώ έχουμε τρία θέματα. Τα ποσοστά 33% και 3,5%. Τα αστυνομικά αυτή στοιχεία οπωσδήποτε θα οδηγήσουν σε πολλές διαφωνίες Πολλοί από αυτούς που συνάντησα μου είπαν να τα μειώσουμε. Άλλοι μου είπαν να τα αυξήσουμε. Ο κάθε διαφορόμενος δηλαδή έχει τη δική του θέση και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των να βρούμε ένα εθνικό στοιχείο που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Αυτό το μέτρο χωρίς να παραβιάζουμε τους ε, κανόνες του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να προσέξουμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά ακριβώς στους νόμους περί ανταγωνισμού. γιατί υπάρχει κίνδυνος οι διαπραγματεύτικέ αυτές ομάδες να είναι ιδιαίτερα ισχυρέ εις βάρος των μικρών παραγωγών. Ένα άλλο θέμα είναι η <clears throat> προστασία της δομής συνεταιρισμών που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Εξαιρούνται βέβαια από το κείμενο, αλλά καταλαβαίνω ότι ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να το διευκρινίσουν καλύτερα το σημείο, αλλά δεν θα είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα μπορούμε να δούμε και τις χώρες που έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής γάλακτος, όπου δεν θα ωφεληθούν από αυτά τα αριθμικά στοιχεία. Να εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο μπορεί να βρεθεί και μια λύση για αυτές. Οργανώσεις των παραγωγών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα ποσοστά και το καθεστώς των συνεταιρισμών. Όσον αφορά τη διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργία των ε, κρατικών αυτών οργανώσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασίζονται βέβαια, σύμφωνα με την πρόταση, σε αυτό που υπάρχει στον τομέα των οπορικευτικών. Αλλά δεν θα έχουν την ίδια όσον αφορά την ε, κατανομή της αγοράς και τον καθορισμό των τιμών. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί κάπως. Δεν θέλω παρά αυτά να πάω πέρα από αυτό που προτείνει η Κομισιόν για το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή. Διαφάνεια. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί είναι κάτι που το συζητάνε πολύ, όταν τους αρέσει και όταν δεν τους στεριάζει το γνώουνε. Μια από τις επιτυχίες, ακόμα ιδίω όταν δεν έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων, και εγώ δεν θέλω να επιστρέφω στο σύστημα των ποσοστώσεων, γιατί θυμάμαι τι έγινε το 2008, όπου η αγορά ελέγχεται από τους ε, παραγωγούς, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχεται το γάλα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια μορφή μηνιαίας παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην Κομισιόν για να ξέρουμε τι παράγουν η παραγωγή στα κράτη-μέλη, ποια είναι η προσφορά, ποια είναι η ζήτηση, γιατί αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ένα ισχυρό σύστημα, για να είμαστε καλά ενημεροί. Αυτό θα είναι καλό και για να καταλάβουμε την κατάσταση στην αγορά και να έχουμε πλήρη επίγνωση των μηνυμάτων που αποστέλει αυτή και να μπορούμε και να αντιδράσουμε. όλοι μπορούν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι αυτό το τμήμα της πρότασης είναι πολύ θετικό. Και εφόσον δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα, περιτά, ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε ένα σύστημα με το οποίο θα μαζεύουμε τα στοιχεία σε κάποιο κεντρικό σημείο και θα μπορούμε να αντιδρούμε έτσι γρήγορα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι ορισμένε από τι οργανώσει με τι οποίε συναντήθηκα μου ζήτησαν να ε, συζητήσουμε το λεγόμενο soft landing, την απαλή προσγείωση δηλαδή, για την οποία πολλοί συζητούσαν στο παρελθόν όταν συζητάμε για την ε, επάψη του συστήματος ε, ποσοστώσεων και τη μετάβαση σε ένα άλλο σύστημα. Θα ακούσω προσεκτικά αυτά που έχουν να πούν οι σκιώδεις ηγητές και τα μέλη της Επιτροπής εδώ για αυτό το θέμα. Σε γενικέ γραμμέ θα πρέπει νομίζω να επιμείνουμε στις προτάσεις όσες έχουν και να μην ανοίξουμε το κουτί της πανδόλας, γιατί καμιά φορά άμα ανοίξει το κουτί της πανδόλας δεν ξέρουμε τι θα βγει από εκεί και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι όλοι ανησυχούν να πετύχουν ένα σύστημα που θα προστατεύσει και θα ωφελήσει τους δικούς παραγωγούς στο γαλακτοκοκό τομέα εκάστοτε. Θα εξετάσω προσεκτικά και σε λεπτομέρειες όλα τα θέματα που σας προανέφερα και ελπίζω η τελική μου πρόταση να μπορεί να υπευληθεί εδώ γύρω στα μέσα Απριλίου. Και προσβλέπω οπωσδήποτε να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών και των μελών της Επιτροπής ε, και θα ακούσω προσεκτικά τις απόψεις αυτές και όπου μπορώ οπωσδήποτε θα προσπαθήσω να βρω μια συμβαστική λύση. Γιατί αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να επιβάλλουμε τη δική μας άποψη για το πώς διαβλέπουμε το μέλλον της, του γαλακτοκομικού κλάδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συζητάμε για τις δυνατότητες επιβίωσης πολλών παραγωγών. Και δεν είναι πάντα εύκολο να, βρεις, να βρούμε μια λύση που να ταιριάζει σε όλους και σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω όμως να πετύχουμε να έχουμε επαρκή ευελιξία για να μπορούμε έτσι να έχουμε τελευταία αναλύσει μια πολιτική που θα εξασφαλίσει δίκαιη επιστροφή για τους παραγωγούς και επεξεργατές του γάλακτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie James. Ευχαριστώ, James. Ευχαριστώ για τη δουλειά σου. Θα αρχίσουμε αμέσως τη συζήτηση. Έχουμε κάποιους εγγεγραμμένους. Η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω κάνοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση κανονισμού που μάλιστα είναι και κριτικές παρατηρήσεις. Η πρώτη ε, αφορά το γεγονός ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο θέλει να προετοιμάσει το μέλλον άνευ ποσοστώσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να εξετάσει ολόκληρο το κλάδο, πράγμα το οποίο δεν το κάνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις επιμένει στις σχέσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και τη βιομηχανία, αυτό είναι ε, το ένα κομμάτι του κλάδου και αφήνει εκτός τη διανομή, δηλαδή το υπόλοιπο κλάδο, όταν σήμερα όλες οι εθνικές αρχές χωρίς εξαίρεση επιβεώνουν ότι το θέμα είναι η διαχείριση που είναι συγκεντρωμένη σε λίγους στο τέλος της αλυσίδας. Οι προτάσει που προτείνονται από αυτό τον κανονισμό βασικά εξυπηρετούν τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλου παραγωγού γάλακτο με δυνατότητε εξαγωγή και που έχουν διάφορε επιλογέ στο επίπεδο ε, παράδοση προ τη βιομηχανία. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου μπορεί λοιπόν, φοβούμε, να οδηγήσει τη συγκέντρωση τη ε, παραγωγή γάλακτο σε μόλι μερικα μερικά κράτη-μέλη που είναι ειδικευμένα και να εξαφανιστεί η παραγωγή στα υπόλοιπα κράτη-μέλη Πράγμα το οποίο είναι αυστηρά απαράδεκτο. Εκτός που δεν ε, διευκολύνει στη διαφοροποίηση που είναι ένα από τα λάβαρα του Επιτρόπου. Εκτός από αυτά τα βασικά, τις βασικές παρατηρήσεις μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε σε θέση σε σχέση με αυτήν την πρόταση να επικαταστήσουμε το σύστημα των ποσοστώσεων που ίσχυσε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα επίσης να κάνω Δύο παρατηρήσεις. Περιορίζω την παρέμβασή μου σε δύο ουσιαστικά ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις συμβάσει Να σας πω ότι ήδη ήρθα σε επαφή με ολόκληρο τον κλάδο για να μπορέσω να συζητήσω και να μιλήσω εξ ονόματός του και ιδιαίτερα στις λέει ότι αυτέ οι συμβάσει πρέπει να είναι υποχρεωτικέ και παρόμοιε για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να μην υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού ανάμεσα στι διάφορε χώρε. Έπειτα, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ οι συμβάσει με συγκεκριμένη ε, τιμή, με ε, τιμαριθμική αναπροσαρμογή και με ενδείξεις για τους όγκους παραγωγής καθώς και για τη διάρκεια των συμβάζων καθώς πρόκειται για έναν τομέα όπου είναι ετήσιες οι αλλαγές. Τι λύσεις λοιπόν θα πρέπει να υποαρουσιάσουμε για αυτούς οι οποίοι δεν ε, έχουν ενταχθεί μέσα στη σύμβαση. Μια δεύτερη παρατήρηση πιο συγκεκριμένη έχει σχέση με τις ε, σχέσεις ανάμεσα στις γεωργικούς συνεταιρισμούς, τους, ε, τις ενώσεις των παραγωγών και τις ε, διαπαγγελματικές ενώσεις. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις απόψεις των διαφόρων οργανώσεων στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα πρότυπο που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για τις ε, διαπαγγελματικέ οργανώσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή ένα πρότυπο τέτοιου τύπου που να εγγυάται μια ειρηνική και παραγωγική συνύπαρξη ανάμεσα στις γεωργικούς συνεταιρισμούς, τους οργανώσεις των παραγωγών και στις διαπαγγελματικές ε, οργανώσεις. Νομίζω λοιπόν, καταλήγοντα ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μα. αν θέλουμε πραγματικά να εγγυηθούμε την βιώσιμη παραγωγή για πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πατραονέβης. Η Ελίζα Γέγκλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας και εγώ διότι μας παρουσίασε πολύ ξεκάθαρα την εν λόγω έκθεση. Η παρέμβαση που μόλις ε, ολοκληρώθηκε δείχνει πως ε, αυτό το μήνυμα ε, προχωρά πολύ περισσότερο από ότι λέει αυτή η έκθεση. Συμφωνώ λοιπόν με τον ε, εισηγητή πως είναι ένα βήμα αυτό, ένα βήμα που θα πρέπει να κάνουμε, αλλά μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Και ήδη το ότι ο επίτροπο μα παρουσίασε μια ανέκθεση είναι μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τον προηγούμενο. Μέχρι στιγμή η έννοια παλή προσγείωση, ομαλή προσγείωση αρκούσε. Τώρα έχουμε και τα σχετικά μέτρα για την εφαρμογή. Μα λένε πάντα ότι το να ε, καταργηθεί το σύστημα των ποσοστώσεων ε, είναι μια απόφαση ήδη λιμένη και ότι εμείς πρέπει να τώρα απλώς να οργανώσουμε την εφαρμογή της. Και αυτή η εφαρμογή, ε, συμφωνώ με τους προϊουλαλίσαντες θα πάρει ακόμα πολύ καιρό και το λέω και εξ ονόματος της Γερμανίας και εξ ονόματος των οργανώσεων με τους οποίες εγώ ήρθα σε επαφή. Φυσικά εννοείται ότι καθένας έχει τα συμφέροντά του και θα ήθελε να προχωρήσουν οι αλλαγές προς τη μία ή την άλλη κατένθεση. Ωστόσο, όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον, νομίζω πως ε, Σήμερα θα πρέπει να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα και θα ήθελα να υποστηρίξουμε το εγγραφό του γιατί τουλάχιστον από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε και το δεύτερο και τρίτο βήμα ώστε τελικά να δούμε πώς θα χειριστούμε τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων γενικότερα. Ή θα μπορούσαμε ίσως και να δούμε τον ε, σχετικό τομέα στην ε, Ελβετία. Ή και να σκεφτούμε την απόλυτη ελευθερία στον τομέα, αν και δεν νομίζω πως κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και είμαι βεβαία ότι ε, θα χρειαστούν ίσως κάποιες τροποποίησεις, αλλά εν γέννη θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσουμε δεχόμενοι ως σημείο το έγγραφο της Κομισιόν και τις προτάσεις του εισηγητήου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ήταν πάρα πολύ καλή η έκθεσή σα. αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, εμπειρίες ε, παραγωγών που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Ε, σύμφωνα με την έκθεση, οι παραγωγοί συνεργάζονται σε κρατικές οργανώσεις, εθνικές οργανώσεις για να προσπαθήσουν τα συμφέροντά τους με τις οργανώσεις πώληση, με τις μεγάλες επιχειρήσεις τις, ε, τις γαλακτοπαραγωγικές στις ε, τέως ε, κομμουνίες χώρες όμως δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή αυτοί οι συνεταιρισμοί και όλα αυτά καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του ε, κομμουνισμού. Για τους παραγωγούς δηλαδή στην Ουγγαρία ο όρος συνεταιρισμός είναι κάτι ανησυχητικό γιατί η ερμηνεία που εδώ δίνεται κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού ήταν κάτι διαφορετικό. Και το μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο πραγματικά, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή. Και μετά τις διαρθρωτικές αλλαγές, μετά την ε, στροφή της ε, πολιτικής, δεν υπήρξε τίποτα που να αντικαταστήσει επιτόπι. Το σημείο κίνησης λοιπόν στις διαπραγματεύσεις είναι τελείως διαφορετικό ε, από αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί στις δυτικές χώρες γιατί για τους παραγωγούς ε, της Ουγγαρίας η ευελιξία, η ελευθερία για συμβάσεις δεν είναι τόσο θετικό όπως είναι σε άλλες χώρες στις πιο παραδοσιακές δηλαδή οικονομίες αγορών στις δημοκρατίες γιατί το σημείο εκείνης της δημοκρατίας είναι τα συμβαλόμενα μέλη να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Στην Ουγγαρία και σε άλλες ε, κομμουνιστικές χώρες δεν ισχύει αυτό όμως. Όταν ο συγητής σας λέει η μεγάλη ευεκκλησία θα ήταν πάρα πολύ σημαντική να μείνουν υποχρεωτικές συμβάσεις αυτές. Ναι, καλό θα ήταν αν όλοι είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες, αν όλοι ξεκινούσαν από το ίδιο σημείο. Αυτό το σημείο ευελιξία σημαίνει για τους μικρούς παραγωγούς να είναι εκτεθειμένοι, έρμεο του κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω, η κατάσταση με τη συμβάση κλπ. είναι πολύ θετική στις παραδοσιακές χώρες, στις δυτικές χώρες, δημοκρατικές. Σε εμά που δεν έχουμε την παράδοση αυτή, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εξ ονόματος των μικρών και μεσαίων παραγωγών θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Σιγητά, να λάβετε υπόψη στην δική μας διαφορετική δομή, τις δικές μας διαφορετικές εμπειρίες. Και θα ήθελα να καλέσω και τις Ουγγρικές Οργανώσεις Παραγωγών να σας διαβιβάσουν αυτές τις πληροφορίες. Και ευχαρίστω να σας καλέσω στη χώρα μου να δείτε επιτόπου τι γίνεται και να συζητήσετε εκεί με τους παραγωγούς για να δείτε πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μορβάη. Τώρα ο κύριος Ταραμπέλα και μετά ο Κώστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω θυμίζοντας ε, από πού ερχόμαστε για να δούμε πού θα προχω... προς τα πού θα προχωρήσουμε. Πριν από το 1984 υπήρξε μια μεγάλη παραγωγή, πολύ πλεονασματικότερη της κατανάλωσης, πράγμα που οδήγησε στο να πληρώνει πάρα πολύ ακριβά η Ευρωπαϊκή Ένωση μια παραγωγή που έπρεπε να αποθηκεύσει και μετά να καταστρέψει. Το ίδιο είχε γίνει και με τα μποροκυπευτικά, όχι μόνο για το γάλα. Και μετά φτάνουμε το... Ε, και εκεί σύγχρησαν τα υποσοστώσεις μέχρι το 2015. Μιλούσαμε τώρα όμως για μια αγορά η οποία δεν τα κατάφερνε και, μέχρι το, και είδαμε το 2009 που μόλις είχε ανακοινωθεί η νέα κατάσταση μέσω της αύξησης ε, του, της ποσός, ποσοστού είδαμε μια μείωση του τιμής που έφτασε ε, από τα 45 στα 18 ευρώ. Ε, λεπτά, συγγνώμη, το λίτρο. Ε, στον παραγωγό. Τώρα, αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, ε, εδώ δεν μιλάμε μόνο βέβαια για μεγάλη ποιότητα που μας έκανε να χάσουμε τμήματα της αγοράς, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει. Αν είναι αυτή η ευελιξία που επιθυμούμε λοιπόν, ναι, γιατί όχι. Αν όμω πρόκειται για ευελιξία τιμών, ε, όπω στην πρώτη πρόταση τη Κομισιόν πρέπει να λάβουμε υπόψη στοιχεία υπολογισμού τη τιμή παρά την ίδια την τιμή και τον καθορισμό τη, θα πω προσοχή. Έτσι δεν διορθώνεται το σημερινό σύστημα. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο σχεδόν ποτέ δεν έχει αναφερθεί. Και εγώ ασχολήθηκα με αυτό το παράδειγμα, είναι το παράδειγμα του Καναδά. Γιατί ο Καναδά ε, λέγανε ναι, οι συμβάσει στην Ελβετία δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά, αλλά έλεγαν ότι ο Καναδά είναι το καλό παράδειγμα. Και εγώ ήρθα σε επαφή με μέλη του Υπουργείου του Καναδικού. Εκεί το σύστημα είναι εξαιρετικά σταθερό. Ξέρετε ποια είναι η τιμή του λίτρου. Είναι 82 σέντ του καναδικού δολαρίου ε, που ισούται με το αμερικανικό. Δηλαδή περίπου 65 σέντ το λίτρο. Και όσοι καταναλώνουν το καναδικό γάλα είναι οι ίδιοι που είναι και εδώ. Δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ε, και εκεί υπάρχει το καναδικό γραφείο γάλακτος που έχει ε, στόχο αποστολή να μεταφέρει από τις φάρμες στους χρήστες του γάλακτος. Και η τιμή επιβαρύνει τον παραγωγό. Είναι 2 σεντ. Τα μεταφορικά. Δηλαδή 59 Σεντ, το λίτρο είναι καθαρά για τον παραγωγό με πολύ μικρές αλλαγές στις ποσότητες και στις τιμές. Βεβαίω ο Καναδάς ε, ασκεί μια πολιτική φορολόγηση στην είσοδο των γαλακτοκομικών προϊόντων που έρχονται από αλλού και έχουν δίκιο. Και βέβαια, ίσω το λέω μόνο για λογαριασμό μου, δεν είχα την ευκαιρία να συμβουλευτώ του συναδέλφου γι' αυτό, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το ε, μεταλλευτούμε και να αμφισβητήσουμε κάποια δόγματα του διεθνού εμπορίου. Δεν μιλάμε σήμερα για τον ΠΟΕ, αλλά να, να αμφισβητήσουμε κάποια δόγματα για το Διεθνέ εμπόριο, για την ε, ανταγωνισμό. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτούνται στον καθρέφτη το πρωί ε, και είναι περήφανοι για αυτά που έχουν καταφέρει στην ενέργεια, για παράδειγμα. Ναι, ο καταναλωτής πληρώνει λιγότερο όλο την ενέργειά του, πιο φθηνά. Οι τηλεπικοινωνίε είναι πιο φθηνέ. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τη ενέργεια ή τηλεπικοινωνία, όπω ή τη τηλεπικοινωνίες όπως η France Telecom για παράδειγμα είναι ικανοποιημένοι καλύτερε οι συνθήκες εργασίας αυτές τι επιχειρήσεις. Και δεν θέλω βέβαια να σα αποσπάσω την προσοχή, αλλά θέλω να ε, κάνω έκκληση για ένα πρότυπο που πέρα από αυτά τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή αντικειμενικοποίηση της τιμής σε κάθε κράτος και του περιθωρίου ε, <coughs> κατάργηση των ποσοστών κτλ. Να δούμε λοιπόν αν ο κύριος Νίκολσον τα βλέπει καλά όλα αυτά. Δηλαδή το δημόσιο χέρι πιο ε, ισχυρό, δηλαδή αν φοβούμε πως αν αναθέσουμε όλη την υπόθεση στα χέρια του ιδιωτικού τομέα δεν θα είναι επιτυχία, λύση. Και πώς θα το κάνουμε, αποθηκεύοντας και πώς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις τιμές με βάση μια δίκαιη ανακατανομή σε κάθε φάση της παραγωγής. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν η τι πιστεύει για όλα αυτά όσον αφορά το, τον κρατικό έλεγχο όλα αυτά. Ναι ή ου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μάρκ Ταραμπέλα. Ε, κυρία Κόστιντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για την πάρα πολύ σημαντική του έκθεση. <coughs> Μου φαίνεται πολύ καλό που αναγνωρίζετε ότι ο γαλακτοκομικό τομέα είναι πάρα πολύ λεπτό τομέα και γι' αυτό αξίζει την προσοχή μα και χρειάζεται και συγκεκριμένε λύσει. Ε, πολύ ενδιαφέρον βρήκα το θέμα της ε, επίλυσης των προβλημάτων τιμών και ε, συνδικαίως ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε στο θέμα της διαφάνειας των τιμών. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά που αναφέρονται. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα όταν μιλάμε και για την ε, διαφάνεια των τιμών να έχουμε κάποιο διακανονιστικό για τις τιμές dumping γιατί ξέρουμε από το παρελθόν ποια είναι η πίεση την οποία υπάρχουν ιδίω οι παραγωγή στις διαπραγματεύσεις ιδίω με μεγάλες ε, <clears throat> αγροδιομηχανικές ε, μονάδες ή τους μεγάλους μεταπολιτές. Ε, και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην παραγωγή γάλακτος στις μειωτούσες περιοχές. Ε, πολλοί παραγωγοί δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν εκείνες τις περιοχές εάν δεν παράγεται γάλα. Και είναι βέβαια λογικό ότι το γάλα στις περιοχές αυτές δεν μπορεί να παράγεται στην ίδια τιμή όπως σε άλλες περιφέρειες. <clears throat> και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν συγκεκριμένε και κατάλληλε λύσεις για τις ορεινές αυτές περιοχές. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επανέλθω στην αρχική πρόταση της δέσμης ποιότητας, όπου υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για τις ορεινές περιοχές και την άμεση εμπορία που αφαιρέθηκαν μετά από το κείμενο. Μου φαίνεται όμως ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο αυτό, ούτως ώστε και όσον αφορά το θέμα την ε, παραγωγή ποιότητας, να δώσουμε στη δυνατότητα και στις περιοχές αυτές να διαθέτουν το προϊόν τους. Ευχαριστώ. Ρέινες. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκολσον για όσα μας είπε και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχήν, τη συζήτηση κατά πόσον θα έχουμε υποχρεωτικές ή μη υποχρεωτικές συμβάσεις. Θα πρέπει να συμφαστούμε την ελευθερία σύμβασης. Ε, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές συμβάσεις, γιατί οπωσδήποτε νομικά αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί. Μετά έχω μια ερώτηση που με έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό όσον αφορά το 3,5% δέσμες ανά Ευρωπαϊκή Ένωση ή 33% ανά κράτος. Πώς ερμηνεύεται αυτό, γιατί λέγεται στην έκθεση ότι θα εξαιρούν τις συνεταιρισμοί. 3,5% από το σύνολο της κοινωνικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένης και της ε, συνεταιριστική ε, ποσόστοση ή όχι, δεν ξέρω. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψεις και θα ήθελα να κάνω να διευκρινιστεί. Να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η βάση από την οποία ξεκινάμε. Και Επίσης το θέμα της διαφάνειας με απασχολεί. Χρειάζεται οπωσδήποτε διαφάνεια για τον έλεγχο, αλλά υπερβολικά πολύ διαφάνεια είναι ει βάρο όλων αυτών που συμμετέχουν στην, ε, στην αγορά. Αν ζητάμε λοιπόν να γίνεται μια παρουσίαση στην ε, Κομισιόν, εντάξει. Από την άλλη μεριά η Κομισιόν όμω θα πρέπει να φροντίσει αυτά τα στοιχεία να μην περάσουν πολύ γλυγορό στην αγορά, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι και οι μεταπολιτές θα έχουν στοιχεία στα χέρια τους για να μπορέσουν να ε, δράσουν εις βάρος ημών των παραγωγών. γιατί όταν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά θα είναι εις βάρος της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών. Και είναι ένα πρόβλημα που είχαμε στο παρελθόν με την ε, διαφάνεια αυτή. Ότι μεγάλες εταιρείε δηλαδή μπορούν πολύ εύκολα να βρουν τα στοιχεία αυτά, ενώ οι μικροί παραγωγοί δεν μπορούν. Δηλαδή καλό είναι ε, να υπάρχει διαφάνεια, αλλά όπως το αλάτι στο φαΐ να μην υπερβάλλουμε. Τρία θέλω να σα πω. Το, το πρώτο είναι κάτι ελευθερία φορά σα πω το σα είδα. Ε, τι έγινε, έπαιζε η Ιταλία, Ιρλανδία στο ράγκμπι το Σάββατο και ήμουν εγώ με τους Γιού μου και με μένα και εμείς ήμασταν με την Ιταλία και μου είπανε πες τα συλληπιτήρια στον πρόεδρό σου γιατί θεωρήσαμε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά η Ιταλία και ευχαριστηθήκαμε γιατί τελικά το τουρνουά των 5-6 κρατών σας πήγε πάρα πολύ τώρα κάτι άλλο. Έχω ήδη απευθύνει στην Κομισιόν για αυτό, αλλά θέλω και να το ξαναπώ, να μας πει θέλει να περνά μια διάταξη στην μεταρρύθμιση αυτή για τα γαλακτοδομικά, ούτως ώστε να έχουμε μια σύμβαση για τις ελάχιστες συνθήκες στα, η παραγωγή, ακόμα και αν τα κράτη-μέλη δεν το κάνουν ό,τι προβλέπει η Κομισιόν υποχρεωτικό. Ήθελα να το ξαναπώ. Τελευταίο κάτι το οποίο για τον Καναδά έφερε ο Μάρκ Ταλαμπέρα. Βεβαίω και είναι κύριο κράτο, αποφασίζει για τη γεωργία του. Και ε, υπάρχουν κάποια θέματα εκεί με την ε, προσφορά και θα ήθελα πάρα πολύ και το Ηνωμένο Βασίλειο να ξεφύγει από το καθεστώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμορφθεί με τον ΠΟΕ, να γίνει σαν τον Καναδά και έτσι να είναι καλύτερα και οι εργαζόμενοι στα γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που υποστηρίζετε την Ιταλία. Ω, ναι, όχι, είναι ενδιαφέρον, είναι ιστορική στιγμή. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία θέλει να πάει με τον Καναδά. Μα εγώ νόμιζα ότι ο Καναδάς θέλει να κόψει τους δεσμούς με την Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια άλλη ιστορική στιγμή φαίνεται. Ε, je crois que c'est intéressant justement qu'on parle du Canada. Νομίζω όμως ότι είναι ενδιαφέρον που μιλάμε για τον Καναδά. Γιατί Δικαίως μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο ε, χειρίζεται την παραγωγή του Καναδά, όπου υπάρχει μια κάποια συνοχή και είναι ένα πρότυπο που λειτουργεί. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και νομίζω πως το έχω πει εδώ ή αλλού, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς διαπραγματεύονται μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ο Καναδάς προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την διάλυση της ε, πολιτικής της στο γάλα και την ε, κατάργηση των ποσοστών. Αν λοιπόν σε αυτή τη λύση είναι τελείως καταστροφικό για τους ε, Καναδούς κτηνοτρόφους αλλά και σε διεθνές επίπεδες γιατί εκεί και οι πολυεθνικές θα κάνουν ό,τι θέλουν. Έχω την εντύπωση ότι τόσο σε διεθνές επίπεδο ε, υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για τους γαλακτοπαραγωγούς που διαφαίνονται με αυτή την κατάσταση του Καναδά. Αλλά θα έλεγα και ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τους παραγωγούς, οργανώνουμε οργανώνεται η προγραμματισμένη εξαφάνιση ενός πολύ μεγάλου αριθμού παραγωγών γάλακτος. Από το 2009 ο αριθμός των παραγωγών που εγκατέλειψαν την παραγωγή δεν ε, αυξάνεται διαρκώς. Είναι πλήρης καταστροφή. Αν απελευθερωθεί η αγορά και είπα το, το σχέδιο αυτό που προτείνει τώρα η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα διότι δεν μπορούμε να... δεν, δεν χειρίζεται τους όγκους. Δεν υπάρχει εγγυημένη βασική τιμή για τους παραγωγούς που ενσωματώνουν την παραγωγή τους. Πώς λοιπόν θα διατηρηθούν αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα παράγουν γάλα τα είναι οι μεγάλες βιομηχανίες, οι κτηνοτρόφοι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να αντισταθούν. Και νομίζω πως είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Πως, γιατί οι συμβάσεις αυτές δεν θα αρκέσουν. Υπήρχαν ούτως ή άλλως. Α, τώρα να μας λένε ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο με βάση τους όγκους είναι γελίο. είναι αυταπάτη να πιστεύει κανεί ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα όταν το 2015 θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Να μην χρειάζεται πια να αποκαλούνται οι ποσοστώσεις. Δεν έχει σημασία αυτό όμω. Το θέμα όμω τη διαχείριση τη παραγωγή ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνολο των κρατών μελών. Δεύτερον, το θέμα της τιμής που πρέπει να καλύπτει το κόστος παραγωγής είναι μια δέσμευση και είναι ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την έκθεση που είχαμε ψηφίσει καταρχήν εδώ στην Γεωργική Επιτροπή και εδώ, θα πρέπει να κρατήσουμε νομίζω μέχρι τέλος. Δεν είναι αποδεκτό το θέμα του κόστους παραγωγής να μην αναφέρεται σαφώς στον κανονισμό. Για τη διαφάνεια, ναι, χρειάζεται διαφάνεια και αυτό το είπαμε και στην Επιτροπή για τη Γεωργία. Για τους μεταποιητές, για τη μεγάλη βιομηχανία, αλλά και για τις αλυσίδες διανομής πρέπει να δώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ποτέ δεν είναι πολύ ε, υπερβολική η διαφάνεια. Γιατί και σήμερα θα μπορούσα να αναφέρω διάφορους βιομηχάνους ε, που κρύβουν τα πραγματικά νούμερα για το κόστος μεταπίσης και κατά τα 20 χρόνια που υπήρχαν οι ποσοστώσεις οι βιομήχανοι είχαν δεχτεί τις τιμές και το λένε διακριτικά Ποτέ δεν έκανα τόσο καλές δουλειές. Γιατί ήταν σίγουροι για τις τιμές και ήταν και σίγουροι για τον όγκο που είχαν στη διάθεσή τους. Να διαχειριστούμε λοιπόν και να εγγυηθούμε τις τιμές δεν είναι καθόλου αντιφατικό με μια βιώσιμη πολιτική για τους παραγωγούς. Ευχαριστούμε. Ζωζέ. Ο κύριος Γιάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τον εισηγητή, την εισηγήτρια γιατί βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση τα γαλακτοκομικά για τη γεωργία της Ευρώπης. Έχω τα Πρώτον μια παρατήρηση. Για μένα οι ποσοστώσεις του γάλακτος ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Θυμάμαι από το 1990 και την επανένωση της Γερμανίας είχαμε πρωτομπεί σε, αυτήν την, σε αυτό το καθεστώ σε αυτή τη ρύθμιση. Το θέμα είναι ότι δίνεται η εντύπωση ότι οι ποσοστώσεις δεν θα πάψουν ποτέ. Μα τότε η γεωργία, γιατί αυτή την ομαλή προσαρμογή να την κάνουν, την ομαλή προσγείωση πώς να την πούμε, Βεβαίω και πρέπει το πρόβλημα να λυθεί σε συνεργασία με τους ε, γεωργούς. Όμως θα πρέπει και εκείνοι να θέλουν να συνεργαστούν. Και έτσι μόνο θα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Τώρα όσον αφορά αυτές τις ποσοστώσεις, ποτέ δεν ήταν πραγματικά ρεαλιστικά προσαρμοσμένες στην αγορά. Να ρίχνω μια ματιά στη δική μου περιφέρεια ο κόσμος εκεί πάντοτε ζητούσε να γίνουν αλλαγές. Ποτέ δεν έγιναν. Γι' αυτό λέω ότι χάθηκαν τόσα χρόνια τόσες ευκαιρίες. Και θέλω να πω για την έκθεση ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν και πολλές εναλλακτικές εδώ η Γεωργία. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα με την Γεωργία. Στη δική μου περιφέρεια έχει κρυθεί αποτυχημένη η ΚΑΠ. Οι τιμές δεν είναι τόσο κακές, αλλά οι εκμεταλλεύσεις έχουν τεράστια προβλήματα. Χρειάζεται αυτό δίκτυο ασφαλείας γιατί έχουμε στρέβλωση στην αγορά οι τιμέ, εάν τυχόν πάρουν την κατηφόρα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βοηθήσει. Τώρα όσον αφορά την παρέμβαση και την αποθήκευση αποθεματοποίηση και εκεί θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις ε, μειονεκτούσε περιοχέ, διότι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουμε και μάλιστα πολύ στα μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Έχουμε το δεύτερο πυλώνα, έχουμε διάφορα προγράμματα στις περιοχές αυτές που τώρα όμως υποφέρουν από κάποια δυνατότητα επιφύλαξης. Γιατί δεν επιτρέπουν να προχωρήσουμε τα εκτατικά προγράμματα. Γι' αυτό θα έλεγα η... ο δεύτερο πυρώνας να ανοίξει και την παραγωγή γάλακτος σε αυτές τις μειοκτούσες περιοχές. Τρίτον, θα ήθελα να κάνω μια σαφή έγκληση όσον αφορά τι οργανώσει των παραγωγών και τι ενώσει του. Χρειαζόμαστε του παραγωγού πρέπει να θέλουν να συνεργαστούν. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε εμείς την, ε, ε, το συνεταιρισμό την Ένωση των Πραγών και τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ως υπηρετορή να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά, να οργανώσουμε τους παραγωγούς και μετά όταν περάσουμε στη πολιτική του Καναδά κλπ. να ξεχάσουμε τι έχω κάνει. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε τη συνοχή, να μην ξεχάσουμε το μέλλον. Αυτές είναι οι επιθυμίες που θέλω να εκφράσω προς τον εισηγητή και ελπίζω κάποιε από αυτές να τις συνστενιστεί. Ε, κατά τα άλλα, να ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή του. Ευχαριστούμε. Κύριε Γιάρ, ο κύριος Όστιν και ο κύριος Γκουτιέρης. Πρέπει να επιταχύνουμε γιατί έχουμε γεμάτη γεμάτη τη διάταξη απόψε. Μάρτιν. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν ε, καθορίσει κανένας ε, κανόνες για την αγορά, δεν βρισκόμαστε στην οδό προς τον, κομμουνισμό, προς τον κομμουνισμό. Μην δεν μπερδεύουμε τα πράγματα αυτά. Άμα εμεί ε, στην πολιτική καορίζουμε κάποιους κανόνες σε μια τόσο ευαίσθητη τομέα, θα πρέπει να διορθώσουμε την υπερβολικά φιλελεύθερη πολιτική των περισμένων ετών. Είναι σημαντικό αυτό. Και δεν θα πρέπει να λέμε ότι επειδή τώρα υπάρχουν πάλι κάποιες τιμές οι οποίες άνοιγε ε, κατά κάποιο τρόπο επαρκήν, όλα τα πράγματα πάνε καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε μια κρίση λόγω υπερπαραγωγής που τελικά ο φορολογούμενος πλήρωνε το ότι εξάγαμε σε τιμές dumping ε, την υπερπαραγωγή αυτή του γάλακτος. Αυτή η κατάσταση μπορούσε να ξαναπαρουσιαστεί. Θα έχουμε πάλι μια κατάσταση λοιπόν. Τα βασικά προβλήματα δεν έχουν επιληθεί συμφωνώ σε ορισμένα σημεία με τον James Nicholson και το έχουμε συζητήσει το θέμα. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε ιδιαίτερα στο θέμα της διαφάνειας. Δεν νομίζω ότι θα βλάψουμε κανέναν να απαιτήσουμε διαφάνεια στην αγορά και θα πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται στην αγορά. Στην πολιτική εμείς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Το ότι έχουμε μια συγκέντρωση στην αγορά γαλακτός που θα ε, αυξηθεί ακόμα περισσότερο γιατί δεν είναι το λιβάδι το αποτελεσματικό στοιχείο πια εκεί που έχουν τις αγελάδες αλλά το πόσο κοντά είναι σε ένα λιμάνι. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε ούτε και με ένα δεύτερο πυλώνα. Και να προσθέσουμε και κάπου 50 ε, ευρώ ας πούμε γιατί δεν μπορούμε να διατηρήσουμε σε αυτές τις περιοχές ε, τις εκεί που τις χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας. Πώς θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τους παραγωγούς στην καθημερινή του ζωή. Δεν νομίζω ότι η πρόεδρος της Κομισιόν δίνει εδώ μια καλή απάντηση. 3,5% των ε, παραγών επιτρέπεται να οργανωθούν. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μετριοπαθές. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή ιδρύεται μια νέα μεγάλη ε, μονάδα επεξεργασία γάλακτος που ενώνει το 5% της αγοράς. Στην Δανία υπάρχει μία οργάνωση αυτή τη στιγμή που επικρατεί σε όλη την αγορά και θα πρέπει να υπάρχουν τρει στο μέλλον. Τι γίνεται μετά οι συνεταιρισμοί. Θα πρέπει να δούμε τι είναι οι συνεταιρισμοί. Ιδίως στην Γερμανία όταν έχουμε κάποιες ε, δομές ε, επιχειρησιακές σε επιχειρήσεις οι οποίες λέγονται με συνεταιρισμένα αλλά ο κάθε συνεταιριστής, ο κάθε παραγωγός δεν έχει καθόλου λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τι λέμε και τι εννοούμε. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ο Καναδάς αναφέρθηκε. Αλλά για να ρίξουμε και ένα βλέμμα προς την Ελβετία. Στην Ελβετία η αγορά είναι αρκετά καθαρή και η κατάσταση των ποσοστώσεων απέτυχε. Εάν λοιπόν δεν το πηγαίνουμε αυτό σε μια τόσο μικρή αγορά, το ότι θα γίνει στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το δούμε δηλαδή και αυτό. Όχι μόνο να κοιτάμε προς τον Καναδά, που καλό παράδειγμα μου φαίνεται, αλλά και εκεί που κάτι τέτοιο προσπάθησαν να το επιβάλλουν και δεν πέτυχαν να μην επαναλαμβάνουμε δηλαδή τα ίδια σφάλματα στην Ευρώπη σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να συζητήσουμε μια τελευταία αναλύση. Ποια θα είναι τα όρια που θα ορίσουμε όσον αφορά την παραγωγή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά ποιο θα καθορίσει η πολιτική, η παραγωγή, οι αγρότες. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω για ποσόσταση, αλλά όταν οριστούν οι ποσότητες θα πρέπει και οι παραγωγοί να έχουν λόγο. Μια απόλυτα απελευθέρωση των αγορών μου φαίνεται ότι θα είναι και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Και μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε. Είχαμε αναθέσει μια μελέτη για τους παραγωγούς, για τους καταναλωτές και βλέπουμε ότι εκεί που ήταν τελείως των αγορά, οι τιμές για τον καταναλωτή ήταν οι πιο ψηλές και για τον παραγωγό οι πιο χαμηλές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε στον Καναδά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ψηλές τιμές για τους παραγωγούς, χαμηλές για τους καταναλωτές. Αυτό ας το έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν. Σέργιο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση που συζητούμε έχει δημιουργήσει σημαντικές προσδοκίες και στο κρατικό τομέα αλλά και στον πρωτογενή τομέα γενικότερα οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα βήμα προς τα εμπρός ο αφορά δηλαδή αλλά και τους ε, ασχολούνται με τα γαλακτοκομικά έχουμε το 2008 τη χρηματιστική κρίση έχουμε το χτύπημα στο χρηματιστήριο οπότε πάρα πολλές επενδύσεις περάσανε ε, στα εμπορεύματα. Ξεκίνησε αυτό στη Νέα Υόρκη, είχαμε όμως ακόμα δύο χρόνια αστάθειας και ε, η κρίση αυτή συνέχισε σαν συγκλονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ε, κατά αυτή τη διατία της κρίσης τελικά είδαμε το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέσα πολιτικής σαν το δίκτυο ασφαλείας. Να και πως φτάσαμε σε αυτή τη συζήτηση, οπότε και εγώ άκουσα το τι γίνεται σχέση με το δίκτυο ασφαλείας, για το κάπως ε, τι χρειάζεται όσον αφορά την παρέμβαση και τη σχετική πολιτική και όπως είπε ο κύριος Ταραμπέλα, θεωρώ ότι δεν είναι φυσικά τέλειος ο κλάδος. Η αγορά των αλλαγωνικών, που δεν είναι καμία αγορά και άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις ατέλειες που πάσχει αυτή η αγορά, Επομένω ε, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την φωνητική θέση των κτηνοτρόφων μας για την αλυσίδα, για τις αρμοδιότητες, για να, είναι για την παραγωγικότητά του, να δώσουν δυνατότητα για αυτές τις συμβάσει που είπαμε, να παρακολουθούμε πιο κοντά τις τιμές, να υπάρχει ονομασία προέλευσης στην ετικατοθεσία και να προχωρήσουμε προς πιο ποιοτική παραγωγή. Να πως θα αλλάξει το τοπίο, αλλά τώρα θέλω κάτι να σα προσθέσω σε αυτό το οποίο συζητήσαμε σήμερα. Πρώτα πρώτα όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις τις συμβατικές. Ό,τι φαίνεται υπάρχουν σημεία προστριβής μεταξύ των συναδέλφων ή της Κομισιόν και ημών και όμω τώρα είναι δύσκολο να κάτσουμε να βρούμε πώς ακριβώς θα δουλέψει πιο καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Όμως, τουλάχιστον, μπορούν να διαλέξουν την ταμείο συμβάσεων τα κρατημέλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί τόσο περισσότερο θα μπορούσαν να έχουν διαπραγματευτική ισχύ αυτή η γεωργοί. Γιατί τώρα έχει κατρακλείσει τιμή και κάτω από, το, από την τιμή, ε, από το κόστος παραγωγής. 4 ή 7% έχει φτάσει σε μερικά μέρη η τιμή του ανέβης εργάς του γάλακτος σε σχέση με το μέσο όρο. Χρειάζεται επομένω πολιτικέ συμβάσει. Αυτό θα βοηθήσει τόσο ώστε να, να εξισορροπηθούν οι ανισότητε και το ίδιο να ισχύσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, θα είναι μια προστεύωση των μέλων. Ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να συμφωνήσουμε για κάποιου περιορισμού, να αποφύγουμε κατάχρηση των ε, των, των διατάξεων να έχουμε ένα 33% μείωση της παραγωγής. Νομίζω ότι είναι εφικτό για τους περισσότερους. Και έτσι, στην αλυσίδα της παραγωγής διατροφικής, να έχει ισχυρή θέση ο παραγωγός. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αφήσαμε τα της ε, εποπτείας της ποιότητας παραγωγής σε κάποιους παραγωγούς και όχι σε κάποια συλλογικά όργανα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τη διαφοροποίηση των χωρών, επομένως ή θα πρέπει να καταργηθεί αυτό το υπάρχον σύστημα ή θα πρέπει να βρούμε το πώς θα κάνουμε μια αποτελεσματική ένωση παραγωγών. Το πιο σωστό επομένως είναι να δώσουμε την άδεια στα κράτη-μέλη να πάνε προς υποχρεωτικότητα των συμβάσεων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν εμπλέγονται την παραγωγή. Το τελευταίο μάλλον θα ήταν πάρα πολύ τολμηρό, αλλά να αποφύγουμε να μην υπάρχει από οποιαδήποτε ρύθμιση λάβουμε καμία προσθεμένη αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων αυτών των βημάτων που γίνεται. Βεβαίως θα πρέπει να, τα κάνουμε τα μέτρα αυτά σαφέστερα, πιο αποτελεσματικά και τελευταίο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει με ευελιξία να ε, φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να τρέχει αυτό το μέτρο το πιο ε, σύντομο δυνατό γιατί διψάνε ένα τέτοιο μέτρο η παραγωγή. Κύριε Σμιθ, κύριε Πρόεδρε, έχω ένα δύο πράγματα να σας πω. Ε, όχι πολλά, γιατί με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Πάρα πολλά θαύμαστα, άξιο θαύμαστα έχει εδώ η Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι επενετή προσπάθεια να μπορέσει να μπει στην χώρα των θαυμάτων σαν την Ελίγη, στη χώρα των γαλακτοκομικών και να τα ρυθμίσει τα προβλήματα. Ε, έχουμε εδώ θέματα που έχουν ανακύψει όμω από την Κομισιόν, γιατί στην αρχή το, το κείμενο θεώρησα ότι σημαίνει πως θα είναι υποχρεωτική η ρύθμιση όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα όμω έχει γίνει εθελουσία, υπάρχει δικαίωμα αυτοεξαίρεση κλπ. Για μένα αυτό θα σημαίνει πισωγύρισμα. Ε, αυτό το να είναι υποχρεωτικά δεν σημαίνει ότι μία ρύθμιση θα αφορά τους όλους. Απλώς ξέρω ως δικαιώστη ότι, υπάρχει ανισορροπία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Και άρα θα πρέπει να γίνουν πολιτικά για τον παράγωγο μόνο μέρο. Κάτι από την Κομισιόν που φαίνεται, μου για εμένα προφανέ, αλλά τίποτα δεν είναι προφανέ εδώ. Μόλι έχουν εκτελεστεί οι συμβάσει, μετά αμέσω μετά μπορεί ε, με τα μεταφορεύσει, α πούμε, να συνάψει άλλη σύμβαση διαδοχική. Για μένα η απάντηση είναι καταφατική προφανώς, αλλά δεν είναι αυτονόητη. Ευχαριστώ τον πρόεδρος, Καπούλα σάντους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εξ ονόματο τη Συστηλιστική Ομάδα ήδη μίλησε ο μας μα εισηγητή που είναι ο Μάρκ Ταραμπέλα, αλλά ήθελα και εγώ να εκφράσω τη δική μου άποψη για το θέμα. Καταρχήν, θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο Γιάρ, γιατί πιστεύω ότι το θέμα του τέλου του καθεστώτο των ποσοστώσεων δεν είναι τόσο προφανή και ε, Διαδικασίε όσο θέλει να μα κάνει να πιστέψουμε. Γιατί έχουμε μια κοινή πολιτική στην Ευρώπη, όλοι το επιθυμούμε αυτό και θέλουμε επίση να διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητε των παραγωγικών ε, περιοχών που έχουν η καθεμία τα δικά τη προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι αναπότρεπτο το τέλο του καθεστώτος των ποσοστών όπω έχει αποφασιστεί, πιστεύω πω υπάρχουν θετικέ επιτυχίες στο έγγραφο που μα παρουσιάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι η Κομισιόν και το η ομάδα υψηλού επίπεδου έδωσε μεγάλη έμφαση στις συμβατικές σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή και τη βιομηχανία. Για κατά την άποψή μου, τα βασικά προβλήματα δεν τίθεται εδώ. Ε, το πρόβλημα είναι όντως η εμπορευματοποίηση, η διανομή των μεγάλων παραγωγών αυτών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα μου θα ήθελα να θυμίσω ότι η σχέση ανάμεσα στους παραγωγούς και τη βιομηχανία, το 75% της παραγωγής είναι, γίνεται από τους συνεταιρισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί η έμφαση που θα πρέπει να δοθεί. Είναι το θέμα οι σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή και την βιομηχανία και τις μεγάλες ε, εταιρείε διανομής, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ βασικά. Δύο επαγγελματικέ λοιπόν οργανώσεις και με το maximum διαφάνειας βεβαίω. Ευχαριστώ. Τέλος τη συζήτηση με τον κύριο Σεγκερέσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχετε δει την έρευνα για τα επίπεδα ζήτησης και προσφοράς που προβλέπονται για το 2015 και ποια είναι η στάση των παραγωγών προς αυτό όσον αφορά το επίπεδο παραγωγής. Θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή τους είναι υπέρ αυτή τη ανάπτυξη. Για αυτού του είδου η παραγωγή δεν είναι εύκολη και εδώ οι απόψει ενδιαφέρουν. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είμαι εγώ σκιώδης για την πολιτική μου ομάδα και μέχρι σήμερα έχουμε ενημερωθεί όσον αφορά αυτή την εισήγηση όλα πήγαν καλά, έχω κάποιες παρατηρήσεις όμως. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να πάμε σε μια κοινή ανάλυση και να σταθούμε στο ότι το γάλα είναι ένα προϊόν το οποίο είναι αντικείμενο της ενιαίας αγοράς. Ένα αντικείμενο δηλαδή το οποίο κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Και ε, αυτό γίνεται προς πάσα κατεύθυνση παντού. Επομένως, το να έχουμε μια κοινή πολιτική και ισχυρή για το γάλα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ποσοστώσεις. πέραν του αν πρέπει να πάψουν ή όχι. Ε, μιλάμε για ένα σύστημα 25 ετών που ασκείται αυτή η οχι μιλαμε για Οπότε συλλογικά έχουμε όλοι ως κράτη αποδεχθεί ότι ο καθένας βάζει στην νομοθεσία το λιθαράκι του. Οπότε και φτάσαμε ε, την τελευταία τώρα δεκαετία στην κατάσταση την οποία όταν λένε δύο ευρωβουλευτέ τη λέξη ποσοστό ή δύο υπουργοί, δεν είναι το ίδιο ποτέ να έχουμε αυτή την εξέλιξη τη αγορά όπω έγινε. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Θα πρέπει επομένω και η νομοθεσία να ακολουθήσει, γιατί έχουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ με τη ποσόστοση τη Δανία. Ε, έλεγε η κυρία Φίσορμπολ ότι είναι κάτι σαν φόρο του νέου ιερούς και την άλλη μεριά έχουμε ε, ε, τελείως χαρακτήρα ποσοστώσεις όπως ε, αυτές που ισχύουν στη Γαλλία επόμενες να το λάβουμε όλο αυτό γιατί τώρα το θέμα δεν είναι να κάτσουμε να ξαναφτιάξουμε μια πολιτική με 25 πρόσωπα θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία να είναι ενιαία για ενιαίο προϊόν το οποίο κυκλοφορεί παντού και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που είναι κλειδί το θέμα της αγοράς διότι έχουμε τη σχέση μεταξύ ε, της επιχείρησης και του παραγωγού, γιατί τώρα υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο εμείς οι πολιτικοί να έχουμε υπόψη, είναι η έννοια της ε, επικράτειας της περιοχής. Γιατί το είναι μόνο η περιοχή που μπορεί σε πολλές περιοχές να βοηθήσει τη οικονομικής, αλλά όμως δεν είναι η ίδια κατάσταση παντού όσον αφορά την απόδοση. Άρα σε μια αγορά σαν την αγορά γάλακτος δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει κάποια δεδομένα τα οποία είναι δεσμευτικά για το μέλλον. Άρα θέλουμε να μην βρεθούμε να προσπαθούμε να διηγηθούμε την απερίμωση ορισμένων περιοχών. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι βάση εδώ είναι οι παραγωγές, η παραγωγή, είπαμε ότι έχουμε το θέμα των συμβάσεων, σύμφωνοι, αλλά είδατε γιατί πρέπει κανεί να είναι σε αυτές τι ρυθμίσεις, ε, γιατί πρέπει να είναι προσεκτικό. Δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια μέτρα τα οποία να ε, μην έχουν κάποια διάρκεια, θα πρέπει να οδηγούν σε επενδύσεις που θα κάνουν η παραγωγή και σε απόδοση αυτών. Ο κόσμος ξέρει τι χρειάζεται. Λοιπόν, θέλουμε να είναι δυνατόν να περάσουν από κάποιον έλεγχο. Γιατί κάποια στιγμή, ιδίω μέσα σε συγκυρία κρίσης, το κράτος θα παρέμβει. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια τα οποία να επιδέχονται αξιοπιστία. Άρα εδώ το θέμα είναι η διανομή και η μεγάλη διανομή γιατί έχουμε εδώ την πίεση επί του γάλακτος που ασκείται εκεί πέρα. αν αυξάνονται τα έξοδά τους, έχουν γίνει στα πράγματα που τελικά δεν μπαίνει το γάλα αυτών λοιπόν που αμφισβητούν τη ρύθμιση. Και οπότε σε πολλές περιπτώσεις ε, πάνε και για μείωση της τιμής χωρίς όμως να μπορούν να αποδείξουν τους λόγους που επικαλούν για τη μείωση της τιμής. Τώρα κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί στο έγγραφο είναι ε, η διαχείριση των ποσοτήτων παραγωγής ποιοτικής. Θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μία σχέση με την προέλευση, το, τον τόπο, ε, αλλιώς θα χαθεί το ποιοτικό στοιχείο, θα πρέπει και αυτή η σύνδεση με αυτές τις μεταβλητές της παραγωγής να καλυφθεί. Ναι, Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ούλραντε και σήμερα από την Κομισιόν, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο για να μας πει και τις απόψεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, διστάζω να πάρω το λόγο, γιατί θα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ όλη μέρα. Αλλά δεν νομίζω αυτό να θέλετε, γιατί έχει και άλλα σοβαρά θέματα στην ημερησία σας διάταξη. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα πιο βασικά. Καταρχήν, να πω στον εισηγητή ότι φυσικά είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία μαζί σας για να περάσουμε από αυτή την διαπραγματευτική διαδικασία. φιλοδοξία μας είναι να έχουμε απόφαση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το καλοκαίρι. Ίσως αυτό να είναι κάπως αισιόδοξο, είναι φιλόδοξο σίγουρα, αλλά είναι και ρεαλιστικό. Θα μπορούσε και να γίνει. Δεύτερον, φυσικά αυτή η πρόταση δεν έρχεται από το πουθενά. Βασίζεται στις προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε στη περίφημη ομάδα υψηλού επίπεδου για το γάλα. Και σε αυτό το πλαίσιο είδαμε ποια ήταν τα όρια μέσα στα οποία μπορούσαμε να κινηθούμε και να υποβάλουμε προτάσεις. Δεν πρόκειται βέβαια να αφήσουμε τελείως ανεξέλεγκτη την αγορά, ούτε είναι μια πρόταση που να θέλει να πάει προς τα πίσω και να ρυθμίσει τα πάντα στην αγορά. Αυτό είναι προφανές. Δεν μιλάμε για το απελευθερωμένο πρότυπο της Νέας Ζηλανδίας, ούτε για την υπερρυθμισμένη αγορά του Καναδά ή της ε, Ελβετίας. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγό ε, γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι το 1994. Εκεί είναι που αφήσαμε την κατάσταση και τους αφήσαμε να πάρουν την αγορά οι Νέο Ζηλανδοί και οι Καναδοί. Κάπως παράξενο. Μιλάμε για ένα γαλακτοκομικό τομέα όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω του κλίματός μας, λόγω των δομών μας και λόγω του ότι έχουμε μια παραγωγή γάλακτος που είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα τα κρατημέλη. Είτε μιλάμε για τα μικρά, τα μεγάλα, νότια, βόρεια, δυτικά, ανατολικά. Μιλάμε για κάτι που είναι κρίσιμο στοιχείο στην πολιτική μας. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο τομέας αυτό θα έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικό από τη μία πλευρά, αλλά και να μπορεί να επωφεληθεί αυτού του πλανεκτήματο, αλλά και από την άλλη πλευρά να έχουμε εξισορροπημένη παραγωγή σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών περιοχών, εκεί όπου οι συνθήκες παραγωγής δεν είναι και καλύτερες. Και μπορούμε να πετύχουμε αυτοί στους στόχους, νομίζω, και τους δύο υπόθηκε εδώ και έχουμε ένα δεύτερο πυλώνα όντως που επιτρέπει να υπάρξουν πολλές δυνατότητες για να βοηθηθούν αυτοί οι κτηνοτρόφοι ε, να είναι είτε πιο ανταγωνιστικοί είτε να διατηρήσουν κάποιες συγκεκριμένε συνθήκες. Και στον υπάρχοντα πυλώνα 1 έχουμε το περίφημο 68, το άρθρο 68, μέσω των διατάξεων του οποίου τα κράτη-μέλη μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι σχεδική περίπτωση και να μείνουν μέσα στα όρια το άρθρου 68 και να βοηθήσουν τον κλάδο. Δεν είναι νέο βέβαια ότι το άρθρο 68 δεν θα εξακολουθήσει να ισχύει όπω μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα θα είναι κομμάτι των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση μετά το 2020, ώστε να έχουμε και στο μέλλον τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να διπλασιάσουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες. Ε, τώρα, ετέθησαν κάποιες ειδικέ ερωτήσεις και ήθελα να μιλήσω για αυτές γιατί σίγουρα εδώ θα συνεχιστεί η συζήτηση εδώ σε αυτή την Επιτροπή Γεωργίας για την πρόταση αυτή. Να αναφερθώ λοιπόν σε κάποια από τα ερωτήματα που ετέθησαν. Το ένα ήταν, γιατί δεν καταστήσατε τις συμβάσεις υποχρεωτικές για όλους. Αυτό δεν ήταν δυνατό από ό,τι είδαμε στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επίπεδου, γιατί κάποια κράτη-μέλη, και εξακολουθούν μάλιστα να κατούν την διαστάση, Κάποια κρατημέλη λοιπόν είναι κάθετα κατά της υποχρέωσης ύπαρξης σύμβασης. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε ε, όλη η παραγωγή σε όλα τα κρατημέλη να συμμετέχουν σε αυτές τις συλλογικές συμβάσεις. Δεύτερη ερώτηση ήταν τι θα γίνει σε, κάποια, σε μια περίπτωση όπου ένας παραγωγός βρεθεί σε κάποιο κράτος μέλος όπου ένα κράτος μέλος υπο, ε, ε, αποφασίσει να μην το καταστήσει υποχρεωτικό. Μπορεί να κάνει και αυτό σύμβαση. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί αν το, αν το κράτος μέλος λέει ε, εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από μένα. Και δεν μπορείς εσύ μονομερό να επιμεινεί για να ε, φτιάξει μια τέτοια σύμβαση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει επίση να γνωρίζουμε πω πρόκειται για μια απόπειρα να οθήσουμε τον τομέα τόσο τους παραγωγούς όσο και τις βιομηχανίες, τις μεταπητικές, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από πλευρά των παραγωγών, από πλευρά των μεταποιητών γάλακτος, ώστε να γνωρίζουν τι γίνεται και να μπορούν να παρεμβαίνουν επί τη βάση των σημάτων της αγοράς, να ενημερώνουν τους παραγωγούς και να τους πούνε ναι, εγώ χρειάζομαι μια σύμβαση για συγκεκριμένη ποσότητα και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ώστε να έχω μια σταθερότητα στην προμήθειά μου. Και θα σου δώσω και σένα τη βεβαιότητα σε σχέση με την τιμή που μπορώ να σου δώσω για αυτό το προϊόν, αλλά πρέπει επίσης να έχω την ευελιξία όταν ξεπεράσεις την ποσότητα αυτή να προσαρμόσω και την τιμή. Δηλαδή, στην ουσία τους ενθαρρύνουμε. Ε, ναι, οι συμβάσεις είναι καλές προς το συμφέρον και των διονών και των παραγωγών και των ε, μεταποιητών, αλλά να υπάρχει και μια ευελιξία ώστε να μπορεί να υπάρξει ενημέρωση και προς τους παραγωγούς αλλά και προς τους μεταποιητές για να προσαρμόζονται αναλόγως. Και αυτό έλειπε. Έλειπε το 2008. Ήταν ένα από τους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στα κρίση. Η παραγωγή αύξησαν την παραγωγή του ενώ έπρεπε να τη σταματήσουν. Αν δεν υπήρχε κίνητρο για να τη σταματήσουν, ούτε καμία καθοδήγηση. και δεν υπήρχε όριο για να παραδίδει κανείς την παραγωγή του στο ε, βιομηχανία, ούτε να <coughs> παραδίνει στο συνεταιρισμό και τελικά αύξησαν την παραγωγή ενώ χρειαζόταν να την σταματήσουν τελείως. Τώρα, αν κάποια κράτη με λοιπόν ότι δεν θέλω σύμβαση, νομίζω πως θα βρεθούν στη μειοψηφία. Μιλάμε όμως βασικά για την περίπτωση όπου έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ιδιωτικών ε, μεταπητικών βιομηχανιών, γιατί μετά θα επανέλθω στους συνεταιρισμού. Οι συνεταιρισμοί δεν καλύπτονται ε, αυτοί καθ' αυτοί, γιατί δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση. Υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά όσον αφορά το, η λειτουργία των συνεταιρισμών, γιατί σε ορισμένα οι συνεταιρισμοί και σε αυτό που εγώ γνωρίζω καλύτερα, για να μην σας κρύβω από που προέρχομαι, από εκεί που προερχόταν και πρώην ε, επίτροπος, ε, δηλαδή από τη Δανία, έχουμε συνεταιρισμού και βασικά έχουμε μία, ένα συνεταιρισμό που καλύπτει όλη την παραγωγή γάλακτο. Αυτοί λοιπόν... Τι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι να κάνουν στην αγορά και επίση έτσι μπορούν να δίνουν feedback στου παραγωγού. Ε, όμως το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να πούνε στα μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να σταματήσει αυτές τις παραγωγές γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε εκεί πέρα ε, κάποιες ομάδες παραγωγών οι οποίοι βλέπουν το, τα σύνφα μας εδώ στον ορίζοντα αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε και δεν, υπάρχει μια τέτοια διάταξη επίσης θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους feedback κάποιο είδους ε, διάλογος, ανταπόκριση, αμοιβιότητα ενημέρωση με του παραγωγού. και αυτό θα πρέπει να γίνει με ιδιωτικό τομέα και αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι αν φτάσουμε σε μια νομοθεσία κατά την οποία θα μπορούμε να πούμε ότι τα, η παραγωγή που είναι μέλη της ε, του συνεταιρισμού θα μπορούν να πάνε στο γαλακτοκομείο και να συνεργάζονται εκεί πέρα. Αυτό θα είναι για, προς όφελος των πάντων και έτσι θα αποφύγουμε την κατάσταση όπως έγινε το, 2008 με 2009. Οπότε και η αγορά κατέρευσε. Το 2008-2009 βεβαίω ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση διότι δεν ήταν όλα αυτά αποτέλεσμα του, της διάρθρωσης παραγωγής. Έγινε μια τέτοια κατάψη αγοράς λόγω ζήτησης και αυτό ήταν εξωτερικό σοκ. Ε, αυτά δεν μπορεί να αποκλείσει κανεί. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα σύστημα το, το οποίο να είναι τελείω στεγανό και να μπορεί να αποτρέψει του κλειδονισμού τις αυτού τη οικονομίας. Όμως προσοχή να έχουμε τέλο πάντων κάποιο είδου προληπτική πολιτική. Άρα οι συνεταιρισμοί που σήμερα δεν περπατάνε στην Ευρώπη το, το οποίο ισχύει, ισχύει, δεν είναι αποδοτικές προς την Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει τα μέλη αυτών των συνεταιρισμών να πούνε στα ηγετικά στελέχη τους ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή, βελτίωση και επομένως αυτό θα είναι προς του κλάδου. Να δούνε. Πώς θα γίνουν συγχωνεύσεις, εξαγωγερές τέτοιων συνεταιρισμών. Για να μπορέσουν να έχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην αγορά θα πρέπει να ενώσουν τι δυνάμει τους τόσο ώστε να αποκτήσουν κάποια ισχύ. Δεν τον πείσουν του και κυρίω στον τομέα τη Λιανική, γιατί ο κλάδο τη Λιανική. εδώ πέρα τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εκμεταλλευτεί τι αδυναμίε όταν έχουμε δηλαδή τόσο μικρά καλακτοκομεία, όταν έχουμε ε, μικρού συνεταιρισμού. Οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί οι μικροί να ενώσουν τους τομείς τους για να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι Από τον εθνικό τομέα επίσης το υπήρχε και ένα άλλο θέμα. Μου φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι για το 3,5% και κατά πόσον αυτό το ποσοστό καλύπτει και τις δύο καταστάσεις εντός ή εκτός ε, συνδεσμού, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα είναι το σύνολο ναι, καλύπτει και το γάλα το οποίο καλύπτει από τα μέλη ενός συνεταιρισμού. Είναι γενική η ρυθμίση, γενική έννοια όσον αφορά το, τη σχέση το, το, τη, μεταξύ αυτονών και του συνόλου της αγοράς. Πάντως, να ολοκληρώσω, αναφέροντάς ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκρισή σας στις προτάσεις μας και εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να είναι πιο τολμηροί και θα ήθελαν πιο δυναμικοί. Δηλαδή να σας πω ότι όταν το 84 ξεκίνησε η ποσοστές τότε στα 10 κράτη-μέλη ήμασταν περίπου ε, στο 1.600.000 παραγωγούς και σήμερα στα ίδια εκείνα 10 κράτη-μέλη έχουμε 220.000 γάλακτο παραβούσε επομένω. Το 84 ξέχνουν οι ποσοστώσεις και από τους τότε 7 εγκατέλειψαν οι 6. Άρα, άρα δεν ισχύει το επιχείρημα ότι οι ποσοστώσεις είναι η λύση. Δεν είναι η λύση απεδείχθη. Δεν βοηθάνε τον παραγωγό. Ίσως επευράδυναν την αναδιάρθρωση, όμως την ύφη την πλήρωσαν εκείνη οι παραγωγοί που θα ήθελαν να επεκταθούν, που, ή που θα... Τόσο θα ήθελαν μέσω της παραγωγής γάλατος να επιβιώσουν και άρα υποστώσεις δεν είναι η απάντηση. Είναι ένα σύστημα το οποίο απέτυχε, διαπιστώθηκε. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαι θέση να επαληθεύσουμε και να επιβιώσουμε ότι αν συνεχίσετε αυτή η συζήτηση όσον αφορά τα υπέρ των ποσοστώσεων είναι κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί τον κλάδο. Εκείνοι, παραγωγή θα πρέπει να επιλέξουν. Να μείνουμε στο σύστημα ή e, να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τις ποσοστώσεις των οποίων απολάβουν και να βγουν από το σύστημα, να βγουν στην αγορά. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν, τώρα έχουμε στο 7% που είναι κάτω από τις ποσοστώσεις, κάτι το οποίο δείχνει ότι το σύστημα δεν αποδίδει, τουλάχιστον ενωσιακά. Βέβαια και κάποια κατημέλη υπάρχει περισσότερη συνέστηση του τι γίνεται. Πρόεδρε, κατόπιν όλων αυτών και εσείς, αλλά και ο εισηγητής, νομίζω ότι καταφέραμε να προχωρήσουμε, να συνεργαστούμε καλά για αυτή την τεχνοκρατική, τεχνική πρόταση. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Όμως προαναφέραμε σε σχέση με αυτή την πρόταση ο πώς δεν θα απαρατηθούμε από την απόπειρα ρύθμιση της αγοράς, το ρόλο μας και ακόμα υπάρχει δυνατότητα να γίνει εξαγορά της παραγωγής. Εις, περίπτωση τα μέτρα που υπάρχουν δεν αποδίδουν. Τα έχουμε σαν ελεκτικό σενάριο. Τι λοιπόν, είπαμε, θέλουμε περισσότερη διαφάνεια. Θέλουμε περισσότερη υπευθυνότητα. Πώς, έχοντας αυτή την Συμβουλευτική Επιτροπή με θεσμικό ρόλο, πάγια λειτουργία και έτσι ενσωπήσουν όλοι τι πραγματικά χρειάζεται ο τομέα και ο κλάδο. Σα ευχαριστούμε κύριε Ούλγαρντ. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα φυσικά. Όλοι θα θέλαμε αυτό το πακέτο μέτρων για το γάλα να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις μας να γίνουν δυνατότερες, πιο ανταγωνιστικές και να αντιμετωπίζουν το σοκ της αγοράς με μέσα που θα τους καθιστούν ικανούς να αποφεύγουν τις μεγάλες μεταβολές της τιμές όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια. Δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολσον και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. James. Ναι, ξέρω πώς πιέζεστε. Γι' αυτό θα είμαι ένα, όσο γίνεται πιο σύντομο να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους καταρχήν για τη συμβολή τους, Κάποιε συντομότερες και κάποιες ε, λιγότερο σύντομε. αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει τη δυσκολία του θέματος, τη δυσκολία του έργου που έχουμε. Να κάνουμε η κυρία Γέγκλε από την αρχή το είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ε, αυτοί που βλέπουν το θέμα και κοιτάνε πώς το εκμεταλλευτούν και άλλοι που το κοιτάνε απλώς ε, και προσέχουν να μην τους ρίξουν. Ο Μάρτιν Χάσλινγκ αναφέρθηκε στην Ελβετία και εδώ υπάρχει ένα ελβετικό στοιχείο σε αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Να μιλήσω με τον Μάρτιν και με την κυρία Γέγκλε. Και αυτό μπαίνει και στα όσα είπε ο Ταραμπέλα για τους Καναδούς. Εγώ δεν έχω εξετάσει αυτό το καναδικό σύστημα σε βάθος, αλλά στην ουσία είναι ένα σύστημα ΑΒ, ποσοστώσεων ΑΒ. Δηλαδή Α είναι υψηλές τιμές και Β είναι χαμηλές τιμές, από ό,τι κατάλαβα. Ίσως πρέπει να το δούμε. Σίγουρα όμω και η Κομισιόν έχει δίκιο που θέλει να κλείσει τη μια συμφωνία μέχρι τον Μάρτιο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πάμε τον Μάρκο στον Καναδά να δούμε ακριβώ πώ λειτουργεί το σύστημα και πόσο αποτελεσματικό είναι. Άρα θα προσπαθήσω να δουλέψω με αυτά που έχω εδώ μπροστά μου. Επίση, αναφέρθηκε και τα προβλήματα των νέων κρατών μελών και μπορώ να πω στη συνάδελφο σίγουρα ότι θα εξετάσω ε, την κατάστασή τους γιατί γνωρίζω και πρόσφατα πήγα στη χώρα της. Ε, αλλά θα πρέπει να πω ότι αν ακούσει κανείς τη σημερινή συζήτηση θα διαπιστώσει ποιες είναι οι δυσκολίες για να βρούμε την μία λύση που θα ταιριάζει σε όλους. Και φυσικά αυτή είναι και η δική μου δυσκολία. Και η κυρία Κώστιγκεν αναφέρθηκε στις ε, ορεινές περιοχές και φυσικά έχει δίκιο και η κυρία ε, Ρέιμες στο 3,5 και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και εδώ υπάρχει δυσκολία και θα πρέπει να το δούμε και με τους σκιώδεις για να βρούμε μια λύση. Και το θέμα της διαφάνειας και πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία στο τέλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η άποψη του κ. Μποβέ για τη συμβάση είναι και επίση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πιστεύω πω ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν μα είπε ότι από το 84 μέχρι σήμερα από του 7 παραγωγού που δούλευαν τότε, οι έξι έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά αυτή. Αλλά αυτό το βλέπουμε και σε άλλους τομείς. Όχι μόνο στο υπαραγωγή γάλακτος. Τώρα, για τον κύριο Γιώνα, να πω, θα πω, ότι ευτυχώ που δεν προσπάθησε που, που είπε συγχαρητήρια και εγώ το είδα με χαρά το παιχνίδι και το ευχαριστήθηκα. Συγχαρητήρια στην Ιταλία. Αλλά έχετε δίκιο ότι αν δεν συνεργαστούν οι κτηνοτρόφοι, δεν θα δουλέψει το σύστημα. Πρέπει λοιπόν κάτι να βρούμε που να θεωρήσουν και εκείνοι ότι θα λειτουργήσει. Και συμφωνώ και με το δίχτυ ασφαλεία. Γιατί όταν η Κομισιόν ε, προσπάθησε να μας ενημερώσει και εμείς πιέζαμε και πιέζαμε η Κομισιόν μπορούσε να έχει αγοράσει πολύ φθηνά και θα το πουλήσει και πάλι με καλά, καλά κέρδη. Με πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν, πόσο λειτουργούσε αυτό το σύστημα και ο κύριος Καπούλα Σάντα και ο κύριος ε, Νταντέ είπαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, τα άκουσα και αυτά με πολύ ενδιαφέρον και άκουσα και την Κομισιόν. Ήδη έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και προσβλέπω στην συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Μια από τις δυσκολίες που έχουμε εδώ είναι ότι ενώ πιέζουμε τους παραγωγούς και τους μεταπιτές να αναλάβουν την ευθύνη για την αγορά, έχουμε ένα στοιχείο εδώ, το μεγάλο στοιχείο, που είναι τα σούπερ μάρκετ βασικά, που ελέγχουν τις τιμές που θα πληρώσουν οι καταναλωτές. Και στη συγκεκριμένη πρόταση δεν μιλάμε τίποτα για αυτούς. Δεν λέμε τίποτα, συγγνώμη, για αυτούς. Οι Γεωργοί, είπατε, δεν ε, σταματήσαν την παραγωγή το 2008 και το 2009. Μα δεν, δεν, δεν έχει κανένα διακόπτη η Αγελάδα, τη πατήσει το κουμπί να σταματήσει να κάνει γάλα, επειδή δεν χρειάζεται το γάλα. Μα αυτό παίρνει καιρό. Χρειάζεται προγραμματισμό και πολλή δουλειά. Και χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία όλων για να υποβάλουμε μια πρόταση που να λειτουργήσει αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, James. Φυσικά και θα επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό αυτό νομοθετικό πακέτο. Περνάμε στο σημείο 5. Παρουσίαση υποπληρές κομισιών του τομέα χείριου κρέατος. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι πως ο τομέας του χείριου κρέατος ε, διανύει κρίση και οι οργανώσεις των κτηνοτρόφων έχουν τονίσει τη σημασία ενός ευρύτατου προγράμματος δράσης ώστε ο τομέας, ε, κοινοτικός τομέας χείριου κρέατος να ξεπεράσει την ε, ζωβούσα κρίση. Επιπλέον επιμένουν για μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για να εγγυηθούμε την παραγωγικότητα του τομέα του χειριού κρέατος και να ενδυναμώσουμε τη δυνατότητά του να, δίνει, να προσφέρει κρέας ποιότητας στον κοινοτικό καταναλωτή και στην παγκόσμια αγορά. Καλέσαμε την Κομισιόν να μας παρουσιάσει την ισχύουσα κατάσταση και τις προτάσεις της, τα μέσα διαχείρισης της αγοράς και άλλα μέτρα για να ξεπεραστεί η κρίση μέσω και μακροπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ, όπω θα γνωρίζετε, έχουν ήδη υποβολή, υποβληθεί μέτρα για την ιδιωτική αποθήκευση του χειρίου κρέατος για να ανακουφιστεί η κατάσταση της αγοράς που είναι πάρα πολύ δύσκολη και το τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας ο Επίτροπος Ντάσιαν Σόλος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανοίξει την δυνατότητα για ιδιωτική αποθήκευση. Θα ζητήσω τώρα από την Κομισιόν, από τον Διευθυντή Ούλγκαρ, να μας ε, παρουσιάσει την κατάσταση. Δεν θα υπάρξει συζήτηση, θα ακούσουμε μόνο την παρουσίαση του κυρίου Ούλγκαρ. Αν επιτέχετε παρατηρήσεις, παρακαλώ τους συναδέλφους να τις γνωστοποιήσουν γραπτώς στη γραμματεία, γιατί δεν έχουμε χρόνο για να ανοίξουμε συζήτηση. Ούλγκαρ, έχεις το λόγο και πάλι. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η κατάσταση μπορεί να συνοψιστεί ως τεχθείς. Στη Γερμανία, όπως ξέρετε, σταθεροποιήθηκε το θέμα της διοξίνης. Έχουμε ορισμένε εκμεταλλεύσει ε, σε καραντίνα ακόμα που ελέγχονται, αλλά το σημαντικό είναι ότι και εκείνε τι εκμεταλλεύσει όπου ε, είναι υποκαραντίνα και όπου αναλύεται το θέμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση κατά την οποία το κρέα που αριχθεί σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις ξεπερνάει τα προβλεπάμενα όρια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό νομίζω. Ότι ακόμα δηλαδή και αν υπάρχει μόλυνση του, ε, των ζωοτροφών, το κρέα αυτό καθ' αυτό ήταν απόλυτα ασφαλές η κατανάλωση. Βέβαια υπήρχαν πάρα πολύ ενδικέ επιπτώσει ε, από το σκάνδαλο αυτό τη διοξίνη και τα ασφαγεία στη Γερμανία μείωσαν μέσα στις τιμές. Τώρα πάντως ε, ξανά επανήλθαν. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε σημαντική αύξηση των τιμών, της τάξης του 10% πάλι. στο οποίο συνέβαλε το άνοιγμα των ιδιωτικών αποθεμάτων. Όπως στην εβδομάδα κατά την οποία αυτό άνοιξε, ε, διαθέστηκαν 37.000 ε, τόνοι. Για τη δεύτερη εβδομάδα δυστυχώ δεν έχω στοιχεία μαζί μου. Για την πρώτη εβδομάδα σας είπα 37.000. Αυτό ήταν ε, μια απόδειξη ότι με την ιδιωτική αυτή αποθήκευση η οδηγή διαγορά κάποια σταθερότητα. Τώρα η διοξίνη βέβαια μειώνεται και ο μηχανισμός ιδιωτικής ε, αποθήκευσης θα βοηθήσει εκείνα τα σφαγεία και εκείνους τους παραγωγούς που δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος τους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν εξεταστεί όλα τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα είναι κατά βάση μια κατάσταση κατά την οποία το κόστος των ζωοτροφών αυξάνεται συνεχώς και μόνο εκείνη η μεγάλη παραγωγή και παραγωγή ζωοτροφών οι οποίοι είχαν, αν θέλετε, τώρα βλέπεις να έχουν μακρά διαρκεία συμβάσεις, μπορούσαν να αποφύγουν για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον την αύξηση αυτή των τιμών των ζωοτροφών. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνοι οι εκτροφείς που πέτυχαν καλύτερα είναι εκείνοι που παράγουν σε μεγάλο ποσοστό τις ζωοτροφές για την εκτροφή στο χειροτροφείο τους. Δεν χρειάζεται να αγοράζουν δηλαδή, τόσο πολύ. Το πρόβλημα είναι εκείνοι οι χειροτρόφοι που αγοράζουν τις ζωοτροφές και οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή λόγω της αύξησης των τιμών. Και έτσι δυστυχώς δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής και να έχουν ένα καλό εισόδημα. Οι τιμές είναι φυσιολογικές θα έλεγα. Δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές μετά τις προσαρμογές που έχουν γίνει. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι αυτή ακριβώς η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και βέβαια και η αύξηση της τιμής ενέργειας. Η αύξηση αυτή επιδεινώνει την κατάσταση για τους εκτροφείς. Δηλαδή υπάρχει πίεση και όσον αφορά το κόστος και όσον αφορά την ε, τιμή πώληση. Και δεν υπάρχει άμεση λύση. Η Κομισιόν προανήγγειλε ότι θα υπάρχει μια σειρά συναντήσεων τους επόμενους μήνες. Η πρώτη συνάντηση αύριο με διευρυμένη συμβουλευτική επιτροπή και έχουμε επίση καλέσει εκπροσωπό από τη γραμματεία σας να συνεδάσει στην συζήτηση αυτή όπου αφενός θα έχουμε εκπροσώπους των κρατών μελών και από την άλλη μεριά θα έχουμε τους συνήθεις εκπροσώπους των ενδιαφερομένων, δηλαδή ραγωγούς, εμπόρους, εκπρόσωπους των σφαγείων, καταναλωτών. Όλοι αυτές συμμετάσχουν στη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με μια σφαιρική παρατήρηση της κατάστασης και βράχη και μακροπρόθεσμα και κατόπιν θα εξετάσουμε τι έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ποια είναι τα μέσα που διαθέτουμε και αυτά που υπάρχουν σήμερα και αυτά όμως που έχουν ζητηθεί στην ανακοίνωση για τη μελλοντική ΚΑΠ. Τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να σταθεροποιήσουμε τις αγορές σε τέτοιες περιπτώσεις. έχουμε μια δεύτερη συνάντηση αρχές Μαρτίου όπου θα έχουμε την παρουσίαση και από κάποιους εμπειρογνώμονες, κάποιους επιστήμονες όσον αφορά το τομέα αυτό. Γιατί και ο τομέα υλοτροφίας και τη εκτροφή πουλερικών που βασίζονται πάρα πολύ στα σιτηρά είναι τομεί στους οποίου δεν είχαμε χρειαστεί μεγάλη παρέμβαση γιατί αυτό διακανονίζονται στο παρελθόν. Είχαμε βέβαια την ειδική αποθήκευση, είχαμε τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, που σήμερα δεν έχει μεγάλο νόημα, γιατί οι διεθνείς τιμές, ε, παραδείγματος χειρίου κρέατος, είναι στο επίπεδο των τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν χάνουμε, αλλά δεν θα κερδίσουμε και τίποτα, γιατί εξαγωγέ χειρίου κράτου αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλέ. Προφανώ είναι γεγονό χρειάζεται κάποια προσαρμογή αυτή τη στιγμή. Η προσαρμογή ή θα γίνει όσον αφορά την προσφορά στον τομέα δηλαδή, της παραγωγής. Το βλέπουμε αυτό σε σχέση με τον αριθμό των ε, χειριδίων ε, και τι θα γίνει με την παραγωγή ή θα πρέπει να γίνει κάτι στην πλευρά των τιμών. Των τιμών δηλαδή της λιανικής Εγώ νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Εάν δεν γίνει κάτι σύντομα όσον αφορά την προσαρμογή, για την πίεση αυτή και τη τιμή και του κόστου, θα υπάρχουν δραματικές αλλαγές. Πολλοί παραγωγοί δεν θα θέλουν ή θα μπορούν να αντέξουν και να συνεχίσουν στην παραγωγή. Ίσως οι τραπεζέ του δεν θα του συνεχίσουν να του υποστηρίζουν. Λοιπόν, εάν ο καταναλωτή θέλει να φάει χείριο κρέας, θα πρέπει να το πληρώσει. Θα πρέπει να πληρώσει υψηλότερη τιμή από την πληρώνει αυτή τη στιγμή. Αλλιώ θα πρέπει να τρώτε πολυρικά ή άλλα κρέατα. Λοιπόν, είναι ε, κατάσταση και διαστρωτικά βράχη πρόθεσμη και διαστρωτικά μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι μια εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και τώρα φέτος έχουμε μια πιο δραματική αν θέλετε εξέλιξη. Έχουμε λίγα μέσα στη διάθεσή μας και το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε κάτι παραπάνω να κάνουμε. Θέλουμε και θα το εξετάσουμε το θέμα. Ένα σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ε, κάπως ε, εμείς ε, πληγώνουμε αυτούς αν θέλετε λόγω των γεννητικά ε, τροποποιημένων οργανισμών γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν φτηνέ ε, ζωοτροφέ που έρχονται από την Νότια Αμερική ή από την Αμερική, τις ΗΠΑ Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν, αλλά δυστυχώ δεν μπορούν να το κάνουν τώρα. Λόγω χρόνου, έλλειψη χρόνου. Παρακαλώ να υποβάλλετε όμως τι ερωτήσεις σας στο γραμματεία. Ευχαριστώ την Γραμματεία για την διαθεσιμότητά τη και για τον τρόπο με τη μέθοδο με την οποία εμπλέκει μονίμω την Επιτροπή μας ε, στη, στα θέματα τα διάφορα. Πάμε στο επόμενο σημείο που αφορά πάντοτε ένα ενημερωτικό σημείο από πλευρά τη Κομισιόν. Πάω γρήγορα γιατί σε λίγο θα πρέπει να δώσουμε το λόγο για του ειδικού μα για αυτό το πολύ σημαντικό σεμινάριο για την ΚΑΠ. Να μας παρουσιάσει λοιπόν η Κομισιόν γρήγορα το νέο μέτρο για τα ίχνη των γενικά τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές, συγγνώμη. Αυτό το σχέδιο έχει ήδη παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη και θα ψηφιστεί στις 8-9 Φεβρουαρίου από την Μόνιμη Επιτροπή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Ε, έχουμε τη διαδικασία επιτροπολογίας με έλεγχο από πλευράς του Κοινοβουλίου μετά από την ψηφοφορία στην Ειδική Επιτροπή θα αποτελέσει τμήμα του ελέγχου από πλευράς Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και θα έχουμε τρεις μήνες. Μιλάει για τη δειγματοληψία και για την εκτέλεση των ελέγχων που θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Και συγκεκριμένα ορίζει το κατόφλι του 0,1% ως το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για να έχει κανείς σημαντικά αποτελέσματα στην ε, δειγματοληψία και τις ελέγχους που γίνονται. Θα δώσω το λόγο στον Γιάρη Μίκο από την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Και εδώ οι συνάδελφοι που θέλουν να αντιδράσουν, τους καλώ να το ζητήσουν από την Γραμματεία. Παρακαλώ, κύριε Μίκο. Thank you very much. Uh, first of all... Uh, let me think. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε το σχέδιο κειμένου μας. Επίσης να σα αναφέρω ότι είναι η πρώτη μου εισήγηση σε αυτή την καινούργια μου θέση, τα καινούργια μου καθήκοντα ή στην διεύθυνση για τα θέματα υγείας που έρχομαι εδώ στη δική σας Επιτροπή, αλλά θα πρέπει με λίγα λόγια να σας εξηγήσω το περιεχόμενο αυτής μας της πρότασης και θα γνωρίζετε ότι ο κλάδος των ζωοτροφών εξαρτάται από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, εξαρτάται πολύ. Ας πούμε, έχουμε όσον αφορά σπόρους 33 εκατομμύρια τόνους το 2008 και 2009 ε, ως επιτοπλίστων από Αργεντινία, Βραζιλία και ΙΠΑ και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ζωοτροφές για την κτηνοτροφία σε τρίτες χώρες. Έχουμε τροποποιημένα και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει όσον αφορά ε, κάποιο συγχρονισμένη έγκριση δικής μας, επομένως υπάρχει ανείχνευση στοιχείων όπως ονομάζεται μια παρουσία σχετικά χαμηλή, προτροποποιημένη σε αυτά τα προϊόντα. επομένω ο στόχο της πρότασής μας είναι να μπορέσουν οι εισαγωγείς να έχουν κάποιο σύστημα και να εισάγουν και εισαγάγουν από εκεί και, και ταυτόχρονα να ισχύει η μηδενική μας ανοχή ως πολιτική που καταρχήν είναι κάτι εύκολο να καταλάβει κανείς αλλά όμως στην πράξη υπάρχουν διάφορες δυσκολίες για τους επισήμους ελέγχους και σήμερα όλα αυτά μας οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλη βεβαιότητα για τους συνελασσομένους στις πολλές δε περιπτώσεις εις τέτοιους κινδύνους οικονομικούς διότι είτε η τιμή των πρώτων υλών έχουν πρόβλημα είτε ο συνελασσόμενος σταματάει να ασχολείται με τις πρώτες ύλες και στην πράξη με την πρότασή μας θέλουμε να εναρμονίσουμε το τι γίνεται με τι συμβάσεις στα κράτη-μέλη, Ούτω ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε οι θεμητέ συνθήκε ανταγωνισμού ή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση θεσπίζονται κάποια πρωτόκολλα για την δειγματοληψία, για τις δοκιμές, για όλα τα κράτη-μέλη, οπότε είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να βρούμε ποιο είναι το ελάχιστο που μπορεί να ανοιχνευτεί από τα, αυτά τα, τα τροποποιημένα και αυτό να γίνεται από τα εργαστήριά μας και με τρόπο που να είναι εναρμονισμένος, να είναι ρεαλιστικός, εφαρμός κλπ. Επομένως αυτό το τεχνικό μηδενικό επίπεδο έτσι το όπως ξέρετε και αντιστοιχεί στο 0,1% και επί τη βάση των όσων έκαναν τα εργαστήριά μας. Ε, τώρα κυρίως μιλούμε τώρα για ζωοτροφές, εκεί όπου εκκρεμεί ακόμα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκεί που έχει εκπνεύσει σχετική αδειοδότηση, εκεί που δεν υπάρχει συμβατότητα με την νομοθεσία για κάποιες ζωοτροφές, τότε... Αυτό πάνε να πει ότι είμαστε παραπάνω από το τεχνικό μηδενικό επίπεδο και αυτή η πρόταση επίσης προβλέπει ότι τα όσα ισχύουν όσον αφορά την ανοίγνωση των ε, των, των, των ε, μεταλλαγμένων ε, παρακολουθείτε. Δηλαδή παρακολουθείτε πάντοτε το επίπεδο των τροπημένων και αν τελικά πάμε παραπάνω από αυτό το επίπεδο τότε αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια και άρα χρειάζεται ειδική απόφαση ακόμα και κατεπίγουσες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε βεβαίω, όπως είπατε πάμε τώρα στην επιτροπολογία για αυτή την απόφαση και είχαμε αυτή την μόνιμη επιτροπή ε, που τώρα τη συζητάει, θα περάσει από εσάς μέσα σε ένα τρίμηνο περίπου. Οπότε με λίγα λόγια αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. E- Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά και μπορούμε γρήγορα γρήγορα να περάσουμε και στο εργαστήριο. Ευχαριστούμε κύριε Μίκο για το, ε, την ενημέρωση. Λοιπόν, εργαστήρι σχετικά με τις συγκεκριμένες πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Να θυμίσω ότι μετά την ακρόαση της 26 Ιανουαρίου με τον εισηγητή Ντες. Είχαμε μια πολύ σημαντική ακρόαση στην αίθουσα της Ολομέλες με όλες τις σημαντικές και αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τη δουλειά μας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και το σημερινό εργαστήρι είναι αφιερωμένο στις τρεις κεντρικές πτυχές της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. στις πληρωμές, μέσα της αγοράς και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και ανάπτυξη της υπαίθρου. Να καλωσορίσω λοιπόν αμέσω τους ειδικού μας, ε, που τους ευχαριστώ, τον Στέφαν Τάγκημαν που είναι ε, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κότιγκεν και πρώην διευθυντή του εμπορίου και της ε, ε, τον κύριο Σατελιέ από το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Οικονομική Έρευνα που είναι πλέον ε, συχνά στην Επιτροπή μας και τον ατήλα Κοφεσόρ από το Πανεπιστήμιο του Βουδαπέστης. Κατα... Προβλέπεται η παρουσίαση από πλευρά των τριών ειδικών. Μάξιμο 20 λεπτά έχουν για την παρουσίασή τους οι τρεις ειδικοί. Σας παρακαλώ να μείνετε στο 20 λεπτό. Και θα έχουμε μετά μία ώρα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Τάγκερμαν πρώτα. Παρακαλώ. <clears throat> Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much first of all for... Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε να εξετάσω την ανακοίνωση της Κομισιόν, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές και που μπόρεσα να συμμεριστώ εδώ τις απόψεις μου. Εξέτασα το κείμενο από τη Σκοπιά μιας καλής αγροτικής παραγωγής. But I now have the being retired and εγώ θα εκφέρω γνώμη εδώ πάνω σε μια πρόταση που εξετάζει αυτή τη στιγμή και δεν είναι ακόμα πολιτική, ώστε θα μιλήσει μόνο για πολιτικές που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Εγώ τώρα όμως είμαι σταξιούχος και μπορώ να μιλήσω και για κάτι που αναπτύσσεται. Και θα το κάνω ανοιχτά, χωρίς διπλωμανικές ε, φιωριτούρε. για να είμαι σαφής. Η ανακοίνωση ορίζει έναν αριθμό σημαντικών ε, προκλήσεων ασφάλεια, τροφιμική, κλιματολογικέ αλλαγέ και ε, δαφυρική ισορροπία. Υπάρχει όμω και μια άλλη πρόκληση, νομίζω, που δεν αναφέρει η ανακοίνωση αυτή, παρόλο αυτή είναι η πραγματική πρόκληση και αφορά την αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον των αμέσων πληρωμών. Αυτές οι πληρωμές αρχικά, όπως ξέρετε όλοι, εισήχθησαν για να ε, υπάρχει ένα αντιστάθμισμα για τους παρόγους, εφόσον υπήρχαν περικοπές των τιμών. Ήταν σημαντικό τότε, δεν μπορούσε να εξεταστεί το θέμα της μεταρρύθμισης της, ε, ε των αμέσων πληρωμών χωρίς να υπάρχει μία, ένα αντιστάθμισμα, μία ε, πληρωμή άμεση προς τους παραγωγούς. Αλλά όταν εισήχθη αυτή η πληρωμή δεν ελήφθη καμία απόφαση όσον αφορά το μέλλον και την εξέλιξη στο μέλλον. Παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Δεν ελέγχθη τι γίνεται εάν δεν χρειάζεται πια αυτό, αυτή η πληρωμή εφόσον θα έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές. Και εγώ βλέπω ότι η ανακοίνωση αυτή της Κομισιόν σε μεγάλο ποσοστό μέσα λέει Ας συμφωνήσουμε να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο αυτές οι άμεσες πληρώμες θα είναι ένα μόνιμο στοιχείο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Και ας συμφωνήσουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν το λέει ρητά, έμεσα όμως η ανακοίνωση το λέει νομίζω ξεκάθαρα κατά τη γνώμη μου αυτό το θέμα του μέλλοντος των άμεσων πληρωμών. Η ανακοίνωση προτείνει μόνο, μόνο πολύ μικρές αλλαγές της πολιτικής. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που προτείνει είναι να αλλάξει η μορφή ενός τμήματο των αμέσων πολιτικών, των αμέσων πληρωμών, συγγνώμη, όσον αφορά την πράσινη στην ιστόσα θα το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που βλέπω εγώ στην ανακοίνωση. Αφενός υπάρχει το κεντρικό σημείο, κεντρικός ρόλος που προβλέπει πάντα η ανακοίνωση για τις άμεσες πληρωμές. Από την άλλη μεριά όμως φοβούμε ότι δεν είναι σαφές γιατί οι άμεσες πληρωμές είναι το μέσο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Δηλαδή με λίγα λόγια, η τροφιμική ασφάλεια δεν απαιτεί πληροφέ, πληρωμές στην Ευρώπη για να μπορέσει η Ευρώπη να συμβάλλει στην ασφάλεια αυτή σε διεθνές επίπεδο. γιατί υπάρχει το πρόβλημα εκείνων που δεν μπορούν να αγοράσουν τρόφιμο γιατί δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Και βέβαια οι άμεσε πληροφορίε στου παραγωγού τη Ευρώπη δεν καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Ούτε μπορούν να συμβάλλουν στην ανάγκη να παράγουν περισσότερα, μεγαλύτερες ποσότητες η παραγωγή, γιατί εάν χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες στην εθνή αγορά, αυξάνουν τιμές. Και αυτό κανονίζεται λοιπόν άμεσα. Και οι τιμές αυξάζονται και οι αυξαμένες τιμές λένε στους παραγωγούς να παράγουν κάτι παραπάνω. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην ε, ΚΑΠ το του και το 80 και οι άμεσες πληρωμές δεν μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ε, κοινοτικής πολιτικής. Εάν ανταγωνιστικότητα σημαίνει η ικανότητα τη... να διατεθούν το τρόφιμα αυτό στην αγορά βάσει της παραγωγικότητας ε, της αγοράς. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους περισσότερα χρήματα και μετά να του επιτρέψουμε να ανταγωνιστούν. Αυτό δεν είναι πραγματική, πραγματικός ανταγωνισμός. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς η παραγωγή βελτιώνεται μέσω της πραγματικής ανταγωνιστικότητας. Αν περάσουμε τώρα στις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, υπάρχουν ε, πολλές απαιτήσει ειδικέ για την εγκατάσταση. Ορισμένοι θέλουν να προωθήσουν την βιοποικιμορφία, άλλοι θέλουν να, να, να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές με τη συλλογή άνθρακα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια απάντηση για όλους. Άρα ο δεύτερος πυλώνας θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα και το ίδιο ισχύει και για την εδαφική ισορροπία. Γιατί ξέρουμε ότι οι διάφορες ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν σημαντικότητα όσον αφορά τη συμβολή της γεωργίας και την δυνατότητα συμβολής της γεωργίας για την οικονομική και κοινωνική ισορροπία των περιοχών αυτών και να υπάρχουν άμεσες πληρωμές ίσες σε όλες τις περιφέρειες δεν υπάρχει επίλυση των προβλημάτων. Δεν είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι η προτινόμενες ε, λύσεις ε, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αναρωτιέται λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος που βλέπει η Κομισιόν για τις άμεσες πληρωμές. Υπάρχει, για να μην το πω πολύ διπλωματικά, υπάρχει μια νέα θεωρία που λέει ότι αυτή η υποστήριξη είναι μια προϋπόθεση για την ικανότητα της ε, κοινοτικής Γεωργίας να παράγει βασικά δημόσια αγαθά αν θέλετε. Δεν ξέρω. Μα πείθει αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Η υποστήριξη του εισοδήματος για λόγους ισότητος με άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα πρέπει να βασίζεται στο εισόδημα των νοικοκυριών, όπως γίνεται συνήθω. σε θέματα τραπεζικά. Και πάλι δεν έχουμε εδώ ένα για τις άμεσες ε, πληρωμές. Και η παραγωγή βασικών δημοσίων αγαθών δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, φαντάζομαι ότι σημαίνει τη διαχείριση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει εδώ απειλή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν καταργούνται τελείως οι άμεσες πληρωμές, δεν θα υπήρχε πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ε, χρήση της γης. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές θα υπήρχε ε, κίνδυνος, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό θα πρέπει να πληρώνονται όλοι οι παραγωγοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι σιγά σιγά λέω ότι αυτές οι άμεσες ε, πληρωμές ανά εκτάριο δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σωστά τις προκλήσεις που υπάρχουν. Και μετά από τα κάπως γενικά αυτά σχόλια θα ήθελα να αναφερθώ σε πιο συγκεκριμένα θέματα, όπως με ζητήθη. Το θέμα των ενεργών παραγωγών. Ξέρετε ότι η ανακοίνωση αναφέρεται στο ότι οι πληρωμές θα πρέπει να δίνονται σε ενεργούς γεωργούς. Εγώ ξέρω ότι είναι ε, Γιώργος, τι θα πει να είναι κανένας ενεργός, δραστήριος, αλλά τι σημαίνει η συνολική αυτή έκφραση. Φαντάζομαι εδώ χρησιμοποιείται για την διάκριση μεταξύ των ε, αγροτικών ε, δραστηριοτήτων και άλλων διαφορετικών χρήσεων της γης. Αν δεν ξέρω αυτό αιτιολογείται, αν πούμε ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων και η χρήση της γης είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, αν κάποιος παραδείγματος ε, κατασκευάζει γήπεδα του γκολφ ή φυτεύει δέντρα γιατί θέλει να κάνει ένα δασάκι και αυτοί δεν χειρίζονται σωστά τη γη δεν προωθούν ε, τους ε, δεν προωθούν τις φυσικούς αυτούς πόρους. Ενεργή γεωργή εν αντιθέσει προς τους απόντες γεωκτήμονες ίσως. Και αυτή είναι μια δυνατότητα να οδεί κανένας. Αλλά δεν λειτουργεί. γιατί οι άμεσες πληρωμές δίνονται ε, στους, ε, στους ε, εκείνους που εκμεταλλεύονται πραγματικά τη γη, αλλά όμως βελτιώνουν έτσι την ε, εκμετάλλευση και το όφελος είναι πάλι στους γεωκτήμονες. Μετά, αν έχουμε τις μικρές ομάδες και τις υπερμεγέθεις. Και εδώ δεν βλέπω να μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα λογικής αλλαγής και πολιτική καπιστικού ορισμού των ενεργών ε, γεωργών. Νομίζω η, η δημόσια ιδέα είναι ότι έχει μια σχέση με τους στόχους που προσπαθούν να επιτευχθούν με την πολιτική αυτή. Έπειτα, υπάρχει ο χειρισμός των μικρών ε, εκμεταλλεύσεων και προτείνεται ένα ειδικό καθεστώ για αυτέ. Έχει νόημα κάτι τέτοιο, αν σκεφτεί κανείς ε, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους. Δεν θα είχε νόημα αν λέγαμε να δώσουμε περισσότερα ας πούμε, αναεκτάριο στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν υπήρχε λόγος για κάτι τέτοιο ούτε θα βοηθούσε αυτό στην προσαρμογή. Αλλά το να μειώσουμε το κόστος των συναλλαγών έχει νόημα. Γιατί αυτό επηρεάζει και την εκμετάλλευση Αλλά όταν κανείς μετά πάει στο επόμενο βήμα και διερωτηθεί πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο μέσω μιας μεγαλύτερης πληρωμής, να καλυφθεί δηλαδή το κόστος της συναλλαγής με μεγαλύτερες πληρωμές, γιατί έτσι δαπανώνται δημόσια χρήματα. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο κόστος της συναλλαγής και τη κέρδος του. Το αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο περιορισμός των διοικητικού κόστους τόσο για την, τον δημόσιο μηχανισμό όσο και για την εκμετάλλευση. Αυτό θα σήμαινε στην ουσία καμία όσον αφορά την ε, την, την συμμόρφωση, την πολλαπλή συμμόρφωση. Οι πληρωμέ θα μπορούσαν να γίνονται μια φορά κάθε πέντε χρόνια ή να δίνονται κάποιο είδου ε, πιστοποιητικά, τα, ε, κάποιοι τα αποκάλεσαν και ομόλογα, Όχι, δεν το προτείνω ω γενικό πρόγραμμα, αλλά για τι μικρές εκμεταλλεύσεις θα μπορούσε κάτι τέτοιο να έχει νόημα και να του επιτρέψει να έχουν μέσα για επενδύσεις για την εκμετάλλευσή του. Επίσης, με, ρωτήθηκε, ε, με ρωτήθηκα ποια θα ήταν ε, η επίπτωση στην ε, πλευρά της προσφοράς. Υπάρχει κάτι το, στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Υπάρχει κάτι το οποίο θα με έκανε εμένα πολύ νευρικό στο πράσινο συστατικό αν ήθελα να υπερασπίσω ένα τέτοιο σύστημα εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο πάνελ επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Διότι, έτσι όπως έχει διατυπωθεί στο ανακοινοθέν, κάποιοι όροι, όπως το ότι θα πρέπει ας πούμε, να έχουν μόνιμα βουσκοτόπια ή ε, αλλαγή εκπεριτροπής των καλλιεργιών. Αυτό το κάνει κανείς ούτως ή άλλως. Αλλά μόνο όταν παράγει. Και ακριβώς αυτό είναι που δεν πρέπει να ζητήσουμε από τους ε, ε, γεωργούς, εάν θέλουμε να μην ε, έχουμε διαφορές στον ΠΟΕ, γιατί αυτό εντάσσεται στο πράσινο κουτί. Αν αυτό το εκτάριο ε, είναι το ίδιο που θα λάβει και το βασικό συστατικό και την ε, πληρωμή, σημαίνει ότι θα απαιτείται να παράγει και άρα δεν θα εμπίπτει στο πράσινο κουτί. βασικό συστατικό τώρα των άμεσων πληρωμών. Ανακατανομία ανάμεσα στα κρατη είναι, κατανοώ το επιχείρημα περί ε, δικαιοσύνης, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν σημαίνει ότι όταν όλοι λαμβάνουν το ίδιο ποσό είναι δίκαιο ή γιατί εγώ είμαι πολύ πιο πλούσιος από ότι ο διπλανός μου ας πούμε ε, δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο όμως αυτό δεν προτείνεται και τώρα όσον αφορά την διάταξη περί δημοσίων αγαθών δεν μπορεί αυτό να αποτελεί τη βάση για την κατανομή των πληρωμών δεν υπάρχει δηλαδή οικονομική λογική εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα εδώ. Το ίδιο δεν σημαίνει και συμβαίνει και με το κάπινγκ. Γιατί ορισμένε εκμεταλλεύσει μπορεί να είναι φτωχέ και άλλε πλούσιε και οι ορισμένοι γεωργοί που φτωχοί και άλλοι πλούσιοι. Αν οι μεγάλοι δεν παίρνουν ένα εκτάριο την ίδια πληρωμή, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι μικρότεροι. Και αυτό σίγουρα δεν είναι προ όφελο τη διορθωτική εξέλιξη. Να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, μιλώντας για το πράσινο στοιχείο. Αυτό είναι το πιο καινοτόμο στοιχείο που θα αντικαταστήσει κάποιο κομμάτι των σημερινών πληρωμών. Θα οδηγούσε σε λιγότερο εισόδημα ανεκμετάλλευση γιατί αυτό δεν καλύπτει το κόστος των έξτρα μέτρων που πρέπει να λάβει κανείς. Οπότε δεν προστίθεται καθαρά, καθαρό εισόδημα. Δεν κατάλαβα ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος ε, που πιστεύετε ότι θα παίξει το πράσινο, το συστατικό θα είναι μια υπέρ ε, συμμόρφωση. Τι είναι, νέα στοιχεία που κανείς δεν τα είχε σκεφτεί και ξαφνικά ξύπνησε και σκέφτηκε ότι πρέπει να περιληφθούν κάποια παραπάνω πράγματα από τη σημερινή συμμόρφωση. Ή πρόκειται για μετακίνηση μέτρων από το δεύτερο πυλώνα στον πρώτο πυλώνα, ώστε τα οικολογικά και περιβαλλοντικά μέτρα να καλύπτονται από αυτό το συγκεκριμένο συστατικό. Και γιατί τότε να πάνε στον πρώτο πυλώνα. Επίσης δεν είμαι βέβαιος αν θα μετακινηθεί και το κονδύλι το αντίστοιχο. Τι θα γίνει με τη σύγχρηματοδότηση. Έχουμε δηλαδή εδώ κάποια ερωτήματα. Αλλά βασικά αυτό που δεν με έχει πείσει Και δεν έχω πιστεί, όπως σας είπα, για το καλύτερη στόχευση των πολιτικών μέσω αυτού του συστατικού, του πράσινου συστατικού. Γιατί τα δημόσια αγαθά είτε είναι πολύ συγκεκριμένη τοποθεσία τους λόγω της φύσης τους ή λόγω του κόστους παραγωγής τους και... και μία ένα καταποκοπήν ποσό για, το ίδιο για όλους δεν θα στοχεύσει πολύ καλά σε αυτά τα μέτρα και οι κυβερνήσει των κρατών μελών θα είναι υποπίεση για να εξασφαλίσουν, να, να, να δουν ακριβώ πόσα χρήματα θα πάρουν από τι Βρυξέλλε. Επίση, δεν θεωρώ πω είναι πιστικό τρόπο για την επιτευξή καλύτερη στόχευση. Υποτίθεται ότι το ανακοινωθέν λέει τι, ποιος είναι ο στόχος και νομίζω αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε η πρόταση αυτή, ότι δηλαδή οι πληρωμές θα γίνουν πιο κατανοητές για τον φορολογούμενο. Εγώ δεν νομίζω πως θα λειτουργήσει ούτε κάτι τέτοιο, γιατί εγώ ως φορολογούμενος βρίσκω μέτρα, τα, τα μέτρα τα οποία βρίσκονται στο δεύτερο πυλώνα πολύ πιο πιστικά από αυτά που είναι στον πρώτο. Τουλάχιστον για μένα προσωπικά δεν είναι πιο κατανοητό ένα τέτοιο μέτρο. Τώρα, οι περιοχές με ιδιαίτερες φυσικούς περιορισμούς και η, θελοντική συνδεδεμένη στήριξη δεν θα μας απασχολεί σήμερα. Θα φτάσω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Ναι, εντοπίζονται σημαντικές προκλήσεις σε αυτή την ανακοίνωση αλλά μόνο περιορισμένες αλλαγές προτείνονται στην κοινή γεωργική πολιτική. Δεν είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση. Τώρα, για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτές τις προκλήσεις στον τομέα ασφάλειας τροφίμων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εγώ θα έλεγα επενδύστε περισσότερο στην καινοτομία και στην έρευνα και την ανάπτυξη. Περισσότερη κατάρτιση, περισσότερη παιδεία, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη λειτουργία των αγορών, χαμηλότερες τιμές γεών. Από αυτά δεν βλέπω πολλά στην ανακοίνωση. Περιβάλλουν κλιματικές αλλαγές που χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα τοπικά, όπως επίσης και η ισορροπία της χρήσης των γεών. Δεν θεωρώ πως το συστατικό το πράσινο είναι καλύτερο ε, εργαλείο για την επίτευξη της ε, καλύτερης στοχοθεσίας. Ε, καλύτερα είναι τα μέτρα στον πυλώνα 2 ε, το κάπινγκ δεν επιτυχάνει την ισότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ε, σωστή η κατανομή μέσω, του, μέσω του κάπινγκ και δεν μπορώ Το έχω εξηγήσει βέβαια και στο έγγραφό μου. Το βασικά μου συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε, είναι ναι, τα δημόσια αγαθά πρέπει να υπάρχουν, η Γεωργία μπορεί να το κάνει, η ανακοίνωση είναι σωστή όταν τονίζει το συγκεκριμένο στοιχείο. Χρειαζόμαστε δημόσια χρήματα, γι' αυτό δεν μπορούν να δώσουν οι αγορές αυτά τα δημόσια αγαθά. Δεν έχω καμία δυσκολία να το καταλάβω αυτό, αλλά όταν θέλει κανείς αυτήν την πολιτική να κάνει μέτρα, καλύτερα είναι να γίνει η πληρωμή αναμονάδα δημοσίου αγαθού και όχι ένα εκτάριο, γιατί το εκτάριο δεν είναι δημόσιο αγαθό. Η συμβολή του εκταρίου στα δημόσια αγαθά μπορεί να μετρηθεί και να ανταμειφθεί. Έχουμε περάσει λοιπόν από την στήριξη της αγοράς στην αποσύνδεση. Επόμενος βήμα θα είναι η στοχοθέτηση και η στοχοθέτηση δεν μπορεί να επιτευχθεί με πληρωμές ένα εκτάριο. Καλύτερα είναι να πληρώνεται η μονάδα δημοσίου αγαθού. Bene, molto bene. Grazie al professor Stefan Tangerman. Σας ευχαριστούμε καθηγητά Tangerman. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Είμαι βέβαιος πως ο Άλμπερ Ντές είναι πολύ ικανοποιημένος για πολλά από αυτά που μας είπατε και Και τώρα να δώσω το λόγο στο δεύτερό μας ειδικό, τον Βίνσεντ Σατελιέ, για 20 λεπτά, μάξιμουμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν έχω την πολυτέλεια που είχε ο προηγούμενος το να είμαι συνταξιούχος, όμως θα τα πούμε κάπως πιο μετρημένα εμείς. Τέλος πάντων, θα είναι και διαφορετικές και σημειώσεις επί των οποίων θα μιλήσω και οπότε θα έχετε πολύ μορφή εδώ στην παρουσία και γι' αυτό θέλω να σας τονίσω ότι Περάσαμε τον Ιανουάριο διαβάζοντας ε, όλα αυτά τα οποία προέβλεπε το Κοινοβούλιο για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Το 1992 ε, ξεκίνησα την διαδρομή μου, τελευταία 18 ετία, ομένως έχω παρακολουθήσει όλες τις αλλαγές στην ΚΑΠ και θα πρέπει να σας πω δύο-τρία πράγματα πριν φτάσουμε στα θέματα της ρύθμισης αγοράς. Πρώτα-πρώτα, ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18 Νοεμβρίου αφορά τα της της οργανώσεις αγοράς και είναι συμβατό διότι δεν θέλει να φέρει σε μήχανη θέση τους εταίρους μας όσον αφορά αυτές τις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Και επομένως γι' αυτό το λόγο αναφέρεται για το ΚΑΠ θα πρέπει να είναι σύμβατη με τις ΚΟΑ. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό οι δασμοί σε μισόμενες χώρες και να ληφθεί υπόψη ο εμπορικός ρόλος των ΚΟΑ. επομενως εδω εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σκοτεινά, λοιπόν, πάρα πολλέ πληροφορίε. Αλλά πρώτα-πρώτα το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά το όποιο θα είναι το ελεκτικό σενάριο εάν κάποια στιγμή ο προπολογισμό συρρυκνωθεί κατά 5 20 οπότε δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πέρα ποια είναι τα κριτήρια που προτείνει η Κομπισιόν Δεύτερο, το κείμενο αυτό παραπέμπει πάρα πολύ σε έναν φιλόδοξο δεύτερο πυλώνα σε αυτή τη διαχείριση των κινδύνων και επομένως το θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτή η συγχρηματοδότηση. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι το η στόχο θέτηση των ενισχύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει αυτού του είδους η υποστήριξη της γεωργίας και πώς αυτό θα είναι ε, κάτι που θα συμβάλλει στο εισόδημα των ε, γεωργών. Επίσης αυτή, ο προσανατολισμός αυτών των ΔΠΟΥ είναι κάτι το αναγκαίο, μια που είναι τόσο ασταθείς οι τιμές, ούτως ώστε το, το, το, το κράτος ενισχύει όχι αυτούς που έχουν ανάγκη, αυτούς που έχουν τις καλύτερες τιμές. Τρίτον, ακόμα και αν το αν όριο για τις ενισχύσεις είναι κάτι περίπλοκο, αυτό θα είναι κάτι θετικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καλύψει τον κοινωνικό σκοπό της, της ΚΑΠ. Παρά το ότι αυτό υπάρχει στην επικουρικότητα, επίση κάτι άλλο το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι επιλέξει, ποιοι ωφελούνται από αυτό το σύστημα γεωκτήμονες στηρίζονται από το κράτος. Αλλά δεν ξέρω εάν αυτό είναι συμβατό με το σύνολο της πολιτικής. Κάτι άλλο, αυτή η καινούρια αρχιτεκτονική θα πρέπει να ξεκαθαριστεί όσον αφορά ιδίω κάποιες μη προνομιούχες ζώνες για τον πρώτο πυλώνα, μετα... και να δούμε σε κάθε φορά τι επιλέγουν, πρώτο ή δεύτερο πυλώνα. Επίσης, επικρίνεται πάρα πολύ η ρύθμιση των αγορών και επίσης έχουμε και όλες αυτές τις ενισχύσεις και επίσης το πώς δίνονται οι άμεσες ενισχύσεις για να δούμε τι θα κάνει αύριο το κράτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν οι γεωργοί όσον αφορά το, το, το ευμετάβολο των τιμών, το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, η αύξηση των η τάση αυξητική και επίση αυτό που γίνεται σε πολλέ αντισώμενε χώρε, Το οποίο μα είναι καλό για την Ευρώπη γιατί έτσι μπορούμε με τι καλύτερε συνθήκε να μειώσουμε τον προστατευτισμό και οι μα μας στι παγκόσμιε τιμέ. επομένω. όταν λέμε αυτό το μεταβόλο αυτό, δεν είναι ομοιογενέ, δεν είναι κάτι ομοιογενέ παντού σε όλου του κλάδου. Έχουμε ας πούμε από τη μία μεριά τα σιτηρά, τα δημητριακά, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και το κρέας που βρίσκεται στην άλλη άκρη του φάσματος. Και όσον αφορά αυτό το, το, μετάβολο των τιμών, ε, τα έχω γράψει εδώ στην έκθεση, αλλά δεν υπάρχει όμως από μεριά από οικονομολόγους μια σύμφωνη γνώμη όσον αφορά το πώς ερμηνεύεται η κατάσταση. Τι οδηγεί περισσότερο διαχρονικά σε αυτή την αλλαγή των τιμών, γιατί φυσικά είναι παραδοσιακά σταθεί οι γεωργικές αγορές, αλλά η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μας οδήγησε πιο κοντά στον ΠΟΕ. Είναι το θέμα επίσης της ε, κάφρα της τιμής των καυσίμων, αλλά έχουμε και την κερδοσκοπία. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το ότι δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη μέσα των οικονομολόγων και επίσης το πώς λειτουργεί ακριβώς η μεταβλητή κερδοσκοπία της αλλαγή των τιμών. Και αυτό κατ' υπάρχει το 2010. Και τελευταία δύο-τρία χρόνια είδαμε να έχει αυξηθεί η σημασία της κερδοσκοπίας. Να, εδώ πέρα αυτό όσο αφορά τη Γαλλία, λέει ο και το άλλο και αφορά ακριβώ την αύξηση του κόστου τη παραγωγή σε μια κατάλληλη γαλλική το 2005 η αύξηση ήταν 20% ε, η 20% μέση αύξηση και μετά είχαμε τι διακυμάνσει ανακλάδο και που τώρα βλέπετε ε, το πόσο μετάβολο ήταν τα γεωργικά εισοδήματα και βλέπετε εδώ πέρα για τα δημητριακά τι έγινε με το εισόδημα μια από το σύστημα των ενισχύσεων δεν προσαρμόστηκε ούτε το 7, ούτε το 8, ούτε το 10 σε σχέση με την τιμή των ε, σιτηρών και οπότε επομένως ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κτηνοτροφία και κατάληξαμε το κάτω να ενισχύει αυτούς που δεν το είχαν ανάγκη. Και δεν ενίσχυσε αυτούς που είχαν πραγματικά ανάγκη. Αυτή είναι η αντίθεση κάποιου που δεν βρίσκεται επιτόπου και τα λέει από καθέδρας του τι χρειάζεται να γίνει. Επομένω, έγινε αυτό το λάθο του διαχείριση δημοσίου χρήματο. Επομένω, το ρίσκο εδώ πέρα είναι παρμεταβλητό, παραγωγή, θέση εμπορία κλπ. Αλλά για εντοπίσουμε αυτό το μετάβολο είναι να έχουμε διαφοροποίηση στη γεωργία, κάτι το οποίο ο δεύτερο πυλώνα το ενθαρρύνει. Όμω αυτό ο πρώτο ε, ε, πυλώνα το φρενάρει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί αυτή η τάση η επιθυμητή για την διαφοροποίηση από τον δεύτερο πυλώνα κυρίω. Πρέπει το πέρα τι γραφικέ παραστάσει να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτέ, ιδίω όσον αφορά τον αυτόνομο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγή. Και αυτό το είπαμε και όσον αφορά το χείριο κρέα, γιατί ισχύει 100% το πιο αυτόνομο σύστημα είναι εκείνα τα συστήματα τα οποία μπορούν να σταθούν όρθια στην κρίση. Και βλέπουμε βέβαια ότι κάθε καινούργια μέρο που θα μπορούσε να επινοηθεί για να έχουμε μια πολιετή διαχείριση μπορεί να περιστύλει αυτό το κίνδυνο των μεταβολών των τιμών. Τώρα όσον αφορά την κρατική πανέμβαση έχουμε τους δασμούς, έχουμε αυτό το κείμενο της Κομισιόν, το οποίο δεν έχει επίκεντρο εμπορικά και τόσο πολύ. Οπότε όσον αφορά αυτούς τους δασμούς και για τη μείωσή τους, αυτό τι, γίνεται. Τι μπορεί να γίνει για την ΚΑΠ. για τον παραγωγό, κέρδος για τον καταναλωτό. Εάν βέβαια υπάρχει η προσφορά. Γιατί υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. να φτάσουμε 85-90% μείωση της ε, προσφοράς και να πάμε εκεί όπως είπαμε όπως στο Βόλιο, όπου οι εξελίξεις αλλού όπως στη Βραζιλία μας οδηγούν στο να καταναλώνουμε περισσότερο, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της προσφοράς. Επίσης έχουμε το, την πολεμή χαρακτήρα όσον αφορά του δασμούς, έχουμε το 50, 54% ε, σε κάποιες χώρες έχουμε αυτή την ιστορική προστασία, στη συνέχεια δε ε, έχουμε τα περίφημα ευαίσθητα προϊόντα που μας ε, οδηγάνε σε μια διαφοροποίηση. Τώρα τι στρατηγική μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρώτα πρώτα δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε στον αφορά της νοβέλ διαστάσεις, οπότε στον ΠΟΕ θερμολάνε και περισσότερο να καλύψουμε τα θέματα τα μη εμπορικά, όπως τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά κλπ. Δεύτερον, οι δασμοί μπορεί να είναι χρήσιμοι σε περιπτώσεις κρίσης. Ε, οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε, ιδίω σε κρίση, να έχουμε κάποιους δασμούς εξωτικού χαρακτήρα για να περιφρουρήσουμε ένα τομέα. Αλλά κάθε κλάδος είναι ευαίσθητο ε, όσον αφορά τους δασμούς, λιγότερο τα δημητριακά, το γάλα, παρά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Δεν είναι και τόσο ευαίσθητος κλάδος γιατί έχουμε ένα 2% εκεί ως αφορά και εισαγωγές και αντιστοίχως όσον αφορά όλα αυτά την ε, ποσοτική διάσταση. Όμως το βόλιο είναι πάρα πολύ ευαίσθητος κλάδος γιατί σε καταστάσεις δύσκολες μπορεί να έχει μεγάλες μειώσεις στους δασμούς. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές, το κείμενο της Κομισιόν ούτε εδώ μας λέει κάτι καινούριο. Αυτό μας οδηγεί στο να υποψιαστούμε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στον ΠΟΕ το 2008 θα συνεχίσουν να ισχύουν. Τώρα, τι στρατηγική μπορεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ε, εξαγωγές, καινοτομία ε, να εκμεταλλευτούμε την πολιτική των επιτοχίων, να έχουμε προσδοκίες ε, για τις, ε, και ελπίδες, κάτι το οποίο μας το γεννά το κείμενο, δηλαδή μεγαλώνει η παγκοσμία αγορά και έχουμε κάποιους ανταγωνιστές όπως την Αυστραλία και άλλες ε, ιστορικά μας ανταγωνίζονται, οι οποίες το έχουν όμως ε, υποχωρήσει και άρα μας αφήνουν χώρο τόσο ώστε να επεκταθούμε εμείς. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι να δεχθούμε ότι οι εξαγωγές επιστροφές είναι δυνατόν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες όσον αφορά μια συγκυρία κρίσης, διότι βεβαίως το ότι δεν θα έχουμε αύριο τέτοιε αρχαιολογικέ επιστροφέ, αυτό δικαιώνει τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει τώρα να κρατήσει χαμηλά τι τιμέ παρέμβαση όσον αφορά την πτυρικότητα των τιμών. Δεν υπάρχει ένα μόνο μέσα, υπάρχουν πολλά μέσα. Τα αποθέματα καταρχήν. Αυτά τα γνωστά αποθέματα ασφάλειας που τα αναφέρουμε συχνά χωρίς να μπορούμε να το ορίσουμε με ακρίβεια. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις φτωχές χώρες που εισαγάγουν σε αντισόμενες χώρες που έχουν δύσκολες, δύσκολους όρους πρόσβασης στους ε, τροφικούς αυτούς Όσον αφορά τώρα τις χώρες όπου η τροφοδότηση είναι πιο εύκολη, είναι ακριβό αυτό. Και όλες οι χώρες του κόσμου δεν θέλουν να αναπτύσσουν τα δικά τους ε, αποθέματα. Λοιπόν, το ένα είναι η στόχη ασφάλειας, η, τα αποθέματα ασφάλειας, συγγνώμη. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι πιο ευέλικτη δημοσιονομικά η ΚΑΠ. Καταλαβαίνω υπάρχουν τεχνικές ε, δυσκολίες, αλλά είναι περίπλοκο. Αν το κοιτάει κανένας απ' έξω, να βλέπει κανένα αυτή την πλήρη ακαμψία του προεμπολισμού σε θέματα που είναι τόσο πτυτικά. Και πάνω σε αυτό δεν κατάλαβα γιατί το κείμενο της Κομισιόν δεν ε, μας δίνει επιχειρήματα που πείθουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τρίτον, και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο, μπορούμε να φανταστούμε ένα σύστημα ε, ε, διακισμάσεων της ε, παραγωγής για βιοκαύσιμα ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά τροφίμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε παραδείγματο χάρη ότι είπα, το 40% του καραβοσίου χρησιμοποιείται στην κατεύθυνση αυτή. Τέλος, όσον αφορά το θέμα της, της πλαισίωσης ε, της κερδοσκοπίας ε, στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντική δυνατότητα εδώ παρέμβαση στις αγορές για το θέμα αυτό. Τώρα, κάτι που αναφέρεται σαν τα υπόλοιπα μέσα για την παρέμβαση της, ε, του κοινού στον, στις γεωργικές μέσα το λεγόμενο safety net, δίκτυο ασφαλεία. Καταρχήν, δεν προβλέπονται νέε μειώσει των δομών για πρώτη φορά. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο τέρμα. Φτάσαμε σε αυτό που επιθυμούσαμε με το 92 να έχουμε δηλαδή ισώσει τις ε, κοινωτικέ τιμές στις διεθνείς τιμές. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να το κρίνουμε αυτό. Μετά, η διατήρηση αυτών των δικτύων ασφαλείας δικαιολογούνται για την αντιμετώπιση εν δυνάμει κρίσεων. Η δημόσια παρέμβαση τη αγορά όμως συνήθως δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματική οικονομικά εάν αυτή η κρίση έχει μαγρά διάκρια. Αυτή η δημόσια παρέμβαση είναι δύσκολη γιατί οι διεθνείς τιμές αυξάνονται και οι τιμές που αποφασίζονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής του που επίσης έχει αυξηθεί. Δηλαδή υπάρχει το δίκτυο ασφαλείας, αλλά η, η κίνηση της λειτουργίας του είναι ε, σπάνια. δεν θα έχουν καμία ή πάρα πολύ μικρή παρέμβαση στα εισοδήματα των παραγών και στην κατανομή του πλούτου, αν θέλετε, μεταξύ αυτών. Πρέπει να δούμε, παραδείγματος, τι γίνεται με τις τιμές παρέμβασης. 101 ευρώ τον τόνο για τα, για τα σιδηρά. Αυτό οφεί ευνοήσουν πολλούς παραγωγούς. Για το κύριο κρέας όμως η τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή και φοβούνται όλοι οι παραγωγοί. Λένε ελπίζω να μην έχουμε καμία σχέση με την τιμή αυτή γιατί τόσο χαμηλή, δεν θα μας οβηλήσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το δίκτυο ασφαλείας, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό. Γιατί οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Μέσα διαχείριση του κινδύνου τώρα. Ε, futures markets. Είναι χρήσιμο το μέσο αυτό για να εξασφαλιστούν και να καθυσυχαστούν οι αγορές αλλά που δεν έχουν καμία επίδραση στην εξέλιξη των τιμών. Είναι ένα μέσο δηλαδή που επιτρέπει να μειώσει τα... τις εχμές χωρίς να έχει καμία επίδραση στις τιμές. Εκτός αυτού, Αυτό δεν έχει επίδραση σε όλες τις τιμές, είναι κυρίως στις τιμές που είναι ε, τυποποιημένες, ιδίως δηλαδή σε κάποιες ε, παραγωγές. Εκτός μπορούμε βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν κοστίζει πολύ το δημόσιο και γι' αυτό είναι δεκτο. Είναι κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά οι παραγωγοί. Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών το γνωρίζουν αλλά που θα χρειαζόταν να, να τους ενημερώσουμε ίσω. Αμυθία κεφάλαια είναι μέσα που δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορεί να βελτιώσουν κάπω στον έλεγχο τη υγεία τη ΚΑΠ, αλλά ίσω είναι καλύτερα προσαρμοσμένα σε ορισμένου τομείς από τις άλλου, όπω τα απορκευτικά. Ε, ασφάλειες κλιματικές, η πολλαπλού κινδύνου, ενδιαφέρον. Στην περίπτωση Γαλλίας, παραδείγματος ανα... προσαρμόστηκαν. Έχουμε την συζήτηση για το άρθρο 68 προηγουμένως. Πράγματι, τα κράτη-μέλη θέλουν να ξέρουν κατά πόσο θα πρέπει να έρθουν τα μέτρα αυτά για να μπορέσουν να προσανατολίσουν την στήριξη σε κάποιους τομείς. Τίθεται και το θέμα της διατησίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Και μετά περνάμε σε κάποια μέσα πιο ε, σύγχρονα κάτι που βλέπω και στα γαλλικά είναι το θέμα την ε, τα προληπτικά μέτρα. Υπάρχουν φορολογικά μέτρα που παρόλες τι προσπάθειες που υπάρχουν και τα μέσα που υπάρχουν ιδίως στη Γαλλία δεν καλούν τους ε, παραγωγούς να ε, αποταμιεύουν προληπτικά και συχνά επενδύουν σε μέσα που δεν οδηγούν σε προσθέμενη αξία. Και το πρόβλημα είναι ότι το 2007-2008 υπήρχε πολύ καλό έτος παραγωγής και τιμών και γι' αυτό η παραγωγοί, για να μην πληρώνουν φόρους δεν ε, αποταμίασαν αλλά επένδυσαν. Λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο καλά και πιο μακριά. Και εδώ τίθεται και το θέμα των ενισχύσεων. Η παραγωγή παίρνουν κάποια ενίσχυση που τη δηλώνουν μετά σε βολογική τους δήλωση. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούν καλύτερα οι παραγωγοί να προσαρμοστούν στην κτητικότητα. Υπάρχει το θέμα της ασφάλεια εισοδήματο. Προσπάθησα να δω τι γίνεται στο Καναδά. Είναι ωφέλιμο αυτό πάντα να κοιτάξουμε τι γίνεται στις Αλλά γιατί να μην χρησιμοποιηθεί ένα μέσο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Το παράρτημα 2 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Μαρικές μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν. Γιατί αυτό μειώνει τους κύριους κινδύνους, κύριους κινδύνους διακύμαση των εισοδημάτων. Το βλέπουμε προφανώς στον Καναδά είναι λοιπόν ένα σύστημα που αξίζει να μελετηθεί. Αυτό βέβαια δεν μπορεί παρά να είναι ένα εκούσιο σύστημα ανάλογο με το ο κάθε κράτος που κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει κατά πόσο θέλει να συνοδεύσει το μέσο αυτό με συν χρηματοδότηση. Βέβαια, όπως λέμε, ο διάβολος είναι στη λεπτομέρεια και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για την ε, ε, ασφάλεια εισοδήματο γιατί κοστίζει πάρα πολύ. Ναι, αλλά μπορούμε να προσαρμόσουμε όμως και τα κριτήρια για να είναι λιγότερο ακριβή και θα πρέπει να δούμε και την ε, διατησία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Και όσα διάβασα από την Κομισιόν δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν διαφορετικές εκμεταλλεύσεις ε, και ερμηνείες ε, εδώ. Για να τελειώσω μέσα στο χρόνο που έχει δοθεί, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τη Γαλλία, παραδείγματο χάρη τις ε, ε, Εγώ ω οικονομολόγο σπάρια ικανοποιήθηκα από την, ε, τα αποδεικτικά σχέδια γιατί θέλουμε τούτο και δεν θέλουμε τ' άλλο. Η Κομισιόν αναφέρεται στη διεύρυνση τη διεθνού αγορά, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην αγορά κλπ. Και Τα καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά στου απολογισμού που γίνεται για τα 25 εφαρμογή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων δεν υπάρχει επιτόπτος κανένα φάκελο που να αναφέρεται στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα και νομίζω ότι οι γαλακτικές ποσοστώσεις είχαν πλεονεκτήματα. Δύο βασικά ε, πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο να ελεγχεται η προσφορά σε χαμηλή τιμή Επίσης υπάρχει μια γεωγραφική κατανομή, δεν είναι ίδιες δηλαδή σε όλα τα κρατημέλη οι ποσοστώσεις αυτές. Επιτρέπει λοιπόν οι ποσοστώσεις να σχετίζονται με τη γη. Οι ποσοστώσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα έλεγα ότι παρόλο που οι γαλακτοκιές ε, ποσοστώσεις στη Γαλλία δεν οδήγησαν στη μείωση των παραγωγών, αλλά είχαν ορισμένα πλεονεκτήματα επιτόπου. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες επικρίσεις, ότι δεν επιτρέπονται με τις ποσοστώσεις να υπάρχει η ιδανική ε, κατανομή των πόρων. Δεύτερον, έχουμε μια τεχνητή αύξηση του κόσμου παραγωγής, γιατί οι ποσοστώσεις μπορούν να απολυθούν. Όχι παντού βέβαια έχω να πω εδώ. Μετά, λέγεται ότι είναι πολύ άγαπτο το σύστημα για να αντιμετωπίσει τις διεθνεί αγορές. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που μπόρεσαν να κατακτήσουν τον κόσμο με συστήματα ποσοστώσεων. Και τέλος, το μέσο των ποσοστώσεων είναι πεπαλαιωμένο, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν είναι πια τυπικό στην πόλη, στην βούληση της ε, του δημοσίου για παρέμβαση. Λοιπόν, υπάρχουν δικαίω θετικά και αρνητικά επιχειρήματα για την ποσόστοση του γάλακτος. Λοιπόν, ποιε είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίε για την κατάργηση των ποσοστώσεων αυτών. Λοιπόν, πρώτον υπάρχει ελπίδα ότι θα αναπτυχθεί η αγορά και θα μπορέσουμε έτσι να ε, ωφεληθούμε από την απόσταση της ωκεανίας στον τομέα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν οι συμβάσεις που είναι χρήσιμες, απαραίτητες, αλλά δεν θα αλλάξουν τα πάντα. Καμιά φορά υπάρχουν ε, ελπίδες που βασίζονται σε συμβάσεις αυτές που ξεπερνούν πολλές φορές την πραγματικότητα. Τρίτον, η τιμή θα μείνει στην ισορροπία προσφορά και ζήτησης και γι' αυτό η διαγραφή των ποσοστώσεων θα αναπτύξει την ζήτηση στην Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι πολλέ χώρε προετοιμάζονται για το τέλο των ποσοστώσεων και πολλοί παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα αύριο να παράγουν περισσότερο γάλα, εάν καταργηθούν οι ποσοστώσει, εφόσον η τιμή του γάλακτος στον, στον, στον ε, τομέα Β θα είναι χαμηλότερη. Επίσης, υπάρχουν δύο θέματα. Το θέμα του κόστου παραγωγής και το κόστος της μεταφοράς του γάλακτος. Για αυτά που άκουσα για τις μενοκτούσε ε, περιοχές είναι σημαντικό. Δηλαδή η ε, κατάργηση των ποσοστώσεων σημαίνει ότι θα συγκεντρώσει γεωγραφικά την προσφορά και θα μπορούσαμε ίσως να διατηρήσουμε τις ποσοστώσεις στις γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές. Και θα πρέπει εδώ να εστιάσουμε έτσι τους δημόσιους πόρους στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του κυρίου Βενσόν Σατελιέ. Φυσικά και ανέφερε πράγματα στα οποία με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και εμείς. Πάμε στην τελευταία παρέμβαση που είναι ο κύριος Ζάμπορ. Παρακαλώ να μείνετε στο χρόνο που σας έχει δοθεί. Έχουμε ήδη πολλούς εγγεγραμμένους να μιλήσουν και φυσικά είναι καλό να μπορέσουν να απαντήσουν οι ειδικοί μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε ένα τέτοιο βήμα υψηλό επίπεδο για να σας εκφράσω τις απόψεις μου για το μέλλον της κοινή πολιτικές, πολιτικής. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες μου στις οθόνες. Good. Μπορείτε να δείτε το περίγραμμα της ε, παρουσίασής μου. Μετά από μια σύντομη εισήγηση, το πρώτο τμήμα της ε, παρουσίασής μας μου θα σας δώσει κάποιες γενικές ε, σκέψεις για την ανακοίνωση της, της Επιτροπής. Το δεύτερο τμήμα αναλύει το ρόλο της ανάπτυξης πέθρου στη μελλοντική και πολιτική και μετά ακολουθούν τα συμπεράσματα. Αρχικά να σας πω ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι υποσυζήτηση για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και για να προετοιμαστεί για την επόμενη πολυετή δημοσιονομική περίοδο. Η Κομισιόν ανέκαθεν έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη διατύπωση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη και δημοσιεύοντα την επίσημη της ανακοίνωση τον περασμένο Νοέμβριο έκανε μια σημαντική συμβολή στην ε, συνεχιζόμενη συζήτηση. Να τονίσω ότι η ανακοίνωση τοποθετείται σε περίπλοκο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον όπου διάφοροι θεσμικοί παράγοντες όπως η Στρατηγική Ευρώπη 2020 ή η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό της μελλοντική κοινή γεωργικής πολιτικής. Η ανακοίνωση εντοπίζει τρεις βασικές προκλήσεις για τη γεωργία στην Ευρώπη ε, και αν κανείς μιλήσει με βιώσιμους όρους μπορεί να το εξονομήσει τις προκλήσεις στην οικονομική, στην περιβαλλοντική και στις κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις ε, θα πρέπει να επιτευχθούν και διάφοροι στόχοι με διάφορες ε, προτάσεις. Έχουμε προκλήσεις, στόχους και προτάσεις εδώ λοιπόν. Και στα επόμενα λεπτά θα αναλύσω την συνοχή ανάμεσα στις προτάσεις και τις ε, προκλήσεις. Ή για να στα πω διαφορετικά, κατά πόσο οι προτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ε, προεντοπισμένες προκλήσεις. Όσον αφορά τη συνοχή των προτάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων, ο στόχος βιώσιμης παραγωγής τροφίμων είναι αυτός που θα πρέπει να επιτευχθεί με διάφορες προτάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, τη σταθερότητα της αγοράς και την, ε, τον κατακαιρματισμό των αλυσίδων παροχής ε, τροφίμων. Εδώ δεν θα μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε για να μην ε, τα ξαναλέω γιατί τα έχουν πει προηγούμενα Τώρα όσον αφορά την συνοχή και την ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, φαίνεται πως η διάταξη περί δημοσίων αγαθών έχει τονιστεί περισσότερο, ενώ η πράσινη ανάπτυξη και οι κλιματικές αλλαγές καθώς και άμβληση των ε, επιπτώσεών τη. δεν ε, αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες προτάσεις. Ωστόσο, οι διατάξεις περί περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών στην Ευρώπη περιλαμβάνουν διάφορες ανεπάρκειες, όπως η ανεπάρκεια της μέτρησης αυτών των αγαθών. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε εκτός από προβλέψεις ε, να κάνουμε για την αξία του τοπίου ή της βιοπικιλότητας στην Ευρώπη και είναι πολύ αμφίβολο να έχουμε την ίδια αξία για τα δημόσια αγαθά, την ίδια μάλλον έννοια για τα δημόσια αγαθά σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά πόσο θα πρέπει να ισχύει η ίδια πολιτική για την παροχή των δημοσίων αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είναι θέμα ποιος θα αξιολογήσει και επί ποιες βάσεις. Ε, κατά πόσο αυτή η πολιτική ήταν ζωστή ή όχι. Επιτυχής μάλλον ή όχι. Και έπειτα, αν δεν μπορεί κανείς να μετρήσει το αποτέλεσμα, είναι πολύ αμφίβολο <laughs> το τι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Όσον αφορά την συνοχή των προτάσεων για την ανταπόκριση των ε, ε, των κοινωνικών και εδαφικών προκλήσεων, να σας πω ότι είναι αρκετά όριστες οι προτάσεις περί ανάπτυξης της υπαίθρου. Περισσότερο ιδέες είναι παρά συγκεκριμένες λύσεις. Οι τρεις βασικοί στόχοι εδώ υποτίθεται ότι θα επιτευχθούν με διάφορες προτάσεις για την στήριξη της απασχόλησης στην υπαίθρο, την ε, βελτίωση της οικονομίας της υπαίθρου και τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση των, συνθήκων για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Αλλά παραμένει σαφές τι ακριβώς προτείνει και είναι τα ακριβή μέτρα, τα συγκεκριμένα μέτρα για να ανταποκριθεί η Κομισιόν στις προκλήσεις αυτές. Φαίνεται ότι η Κομισιόν δεν συνειδητοποιεί, για παράδειγμα, ότι τη διαφορά των δομών των εκμεταλλεύσεων στα νέα κρατημέλη, δηλαδή μεγάλος αριθμός μικρών και μικρότερο των εκμεταλλεύσεων υπάρχει, υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές και αυτές τις εκμεταλλεύσεις είναι απολύτως διαφορετικές από τις μικρές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης των 15. Άρα λοιπόν αυτές οι εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τη σχετική κατηγορία της Ευρώπης των 15. Προκλήσεις για το μέλλον λοιπόν αυτό σημαίνει πως η γεωργική πολιτική θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ε, την ύπαρξη αυτής της κατάστασης και να εφαρμόσει μια διαφοροποιημένη πολιτική. Όχι unisex πολιτική για όλους. Λοιπόν, η Προκλήσεις μεν εντοπίζονται, αλλά οι προτάσεις είναι αόριστες σε, στις περισσότερες φορές. Όπως σα είπα κάποιο προγραμματισμό για την ανακοίνωση τη ε, επιτροπή, να περάσω στο δεύτερο μέρο τη ε, ανακοινώσή μου για το ρόλο τη ανάπτυξη υπαίθρου στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Δεν υπάρχουν αρκετά μηνύματα για την ανάπτυξη υπαίθρου και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά φαίνεται πω ο ρόλο τη ανάπτυξη υπαίθρου στο δεύτερο πυλώνα θα υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ιδέας του πρασινίσματος του πρώτου πυλώνα. Ωστόσο, ο κατάλογος των θεμάτων έχει επεκταθεί και συμπεριλαμβάνεται η καινοτομία και η διαχείριση του κινδύνου, από ό,τι φαίνεται εδώ. Είναι δηλαδή η τμήμα της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήματα που λείπουν. Και αυτά μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε Στι κατηγορίε των μελλοντικών προτεραιοτήτων, την αξιολόγηση των πολιτικών ανάπτυξη πέθρου και ε, τα θέματα τα δημοσιονομικά. Αυτά θα σα τα αναλύσω λεπτομερώς. Όσον αφορά τι μελλοντικέ προτεραιότητε, φαίνεται πως οι επικεφαλίδε πηχούν τη σημερινή δομή της ανάπτυξης της υπαίθρου. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις μελλοντικές προτεραιότητες ανάπτυξης της υπαίθρου, όπως είπαμε. Αλλά υπάρχουν και αμφιβολίες για το πώς θα γίνουν πώς θα, πώς τα κονδύλια σε αυτές τις προτεραιότητες. Με το ισχυρό σύστημα οι πρώτες δύο ε, τίτλοι είναι αυτοί που έχουν την προτεραιότητα, ενώ τα προγράμματα για τη δεύτερη επικεφαλίδα ή το δεύτερο άξονα δεν ε, αντιμετωπίζονται. Είναι απογοητευτικό, για παράδειγμα, ότι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα στις περιοχές της υπαίθρου, δηλαδή η φτώχεια, δεν αναφέρεται καν στο κείμενο να τονίσω ότι η ελάφρυνση της μεγάλης φτώχειας στην Ήπεθρο θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό κλειδί, πολιτική κλειδί στο μέλλον, που στόχο θα έχει την μείωση του χάσματος μεταξύ των εισοδημάτων των αστικών κέντρων και των εισοδημάτων της Υπέθρου, που αυξάνεται εδώ και μερικά χρόνια στην Ευρώπη. Όσον αφορά την αξιολόγηση των πολιτικών για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, έχουν προκύψει διάφορες επικρίσεις σε σχέση με το ισχύον σύστημα αξιολόγηση που βασίζεται στην κοινή παρακολούθηση και κοινό πλαίσιο αξιολόγηση. Και εν μέσω αυτών που επικρίνουν θα πρέπει να τονίσουμε το ότι εδώ πέρα υπάρχει το πρόβλημα το ότι αυτοί οι δείκτες δεν καλύπτουν το τι έγινε. Απλώς λένε τι έγινε στην Ήπεθρο, αλλά όχι το πώς έγινε. Οπότε και χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μία στροφή προς μία αξιολόγηση από τη βάση του αποτελέσματος. Να έχουμε επομένω αξιολογήσεις από τη βάση μετρησίμων στόχων. Και θα πρέπει να υπάρχει feedback των αποτελεσμάτων προς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ε, επίσης, θα πρέπει να βρούμε κάποιο είδου στόχου, είπαμε, ποσοτικά αποτιμητού και θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδου εφαρμογή, ούτω ώστε οι στόχοι τη ΕΕ να συνδέονται με τις γενικότερες ενωσιακές προτεραιότητες για όλες τις πολιτικές και οι στόχοι να βασίζονται στο δόκιμον, το δέον, το εφαρμόσιμο ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το διφυή χαρακτήρα των στόχων τον καλύψουμε να αλλάξει επομένω το σύστημα αξιολόγηση στο, στο μέλλον, λέω. Και έτσι να έχουμε δύο μεθόδους. Την μακροπροσέγγιση και την μικροπροσέγγιση. Information. On the one hand, Οπότε έτσι οι δείκτες της μακροπροσέγγισης να μείνουν ίδιοι, όμως χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει αναθεώρηση των σημερινά χρησιμοποιημένων δικτών για να δούμε τι θα γίνει με τους στόχους των προγραμμάτων. και έτσι να έχουμε κάποιες ε, περιφέρειες που να μελετηθούν ως παραδείγματα για να δούμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε. Και έτσι να δούμε πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να έχουμε όλο το ψηφιδωτό. Τι έγινε, πώς έγινε στην Ήπεθρο στην Ευρώπη. Τώρα το τελευταίο είναι οι προβληματισμοί οι δημισιονομικοί. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρόκειται να περικοπεί στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα διάρθρωση των πόρων ανά κρατός μέλος και ανά πυλώνα. Όμως, το ότι κάποια μέσα από το δεύτερο πυλώνα θα πάμε στον πρώτο πυλώνα, τι πάει να πει. Πάει να πει ότι έτσι θα πάμε σε κάποιον ανασχηματισμό των κονδυλίων των διατηθεμένων. Το οποίο χρειάζεται. Χρειάζεται από τα κράτη-μέλη, μια που η σημερινή κατανομή των κονδυλίων μέλος είναι πάρα πολύ άνηση. Οπότε, βασικά, έχουμε ε, την αναμάσταση των παλαιότερων συμφωνιών που δεν είναι πλέον ρεαλιστικές. Εις δε το κείμενο της ανακοινώσεως αναφέρεται το ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία να είναι καθαρά, σαφή και θα πρέπει αυτό να γίνει από τη βάση των όσων προτείνουν οι εμπειρογνώμονες τη Ένωση. Να βρούμε λοιπόν κάποιου συγκεκριμένου δείκτες και αυτοί να μας εξυπηρετήσουν καλύτερα για να μπορέσουμε να τους συνδυάσουμε με αντικειμενικά κριτήρια. Να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ κατά κεφαλή, το Natura 2000, η έκταση, η χρησιμοποιούμενη για γεωργία και αυτά όλα να λαμβάνει υπόψη τις ε, αηφόρες κατηγορίες. Στην Ευρώπη. Σε σχέση επίσης με αυτούς τους προβληματισμούς μας, θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκαθαριστεί η, ο ρόλος Τη ανάπτυξη τη υπαίθρου. Στα πλαίσια τη γεωργική Πολιτική. θα πρέπει να έχουμε πολιτικές αντίστοιχε. Και θα πρέπει επομένως να υπάρξει μια τέτοια πολιτική. Και όλα αυτά να βελτιωθούν όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και γι' αυτό και εγώ εντόνω, συνιστώ όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα νέο ταμείο. Να έχουμε έτσι περισσότερο αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξη της Πέτρο, Να μειώσουμε τις επικαλύψεις που ισχύουν σήμερα για τα κοινωτικά ταμεία και επίσης έτσι να έχουμε καλύτερο συντονισμό των πολιτικών. Τα σημερινά προγράμματα τα διαχειρίζονται εθνικοί φορείς. Ουδέποτε υπήρξε ενσωμάτωση και ένταξη εις μια ενωσιακή πολιτική και για αυτό θα πρέπει να γίνει μια τέτοια ένταξη στο γενικότερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη της Πέθρου. Ε, τα συμπεράσματα τώρα είναι μάλλον πρόημο για να κάτσουμε και να δούμε τον ρόλο της ή στην ΚΑΠ του μέλλοντος. Όμως, μπορούμε να δούμε τι άλλα συμπεράσματα έχω εξαγάγει. Στο πρώτο μας παρουσίαση σας ετώνησα ότι οι προτάσεις αυτές δεν είναι λεπτομερείς. Εν μέρη μόνο συμβαδίζουν με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Από ό,τι φαίνεται δε, η ΚΑΠ του μέλλοντος θα διέπεται από διάφορε θεσμικέ μεταβλητέ που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Διότι ο ρόλο τη της Πέθρου, από ό,τι φαίνεται, στο δεύτερο πυλώνα είναι υποβαθμισμένο. Άρα πάμε εις μια γενικευμένη υποβάθμιση της πολιτικής ανάπτυξης της Πέθρου. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με το περιβάλλον το οποίο Σοβάκη πρασινίζει τον πρώτο πυλώνα. Άρα στο μέλλον ίσω δεν θα πρέπει να αλλάξουν προτεραιότητε. Όμω, η φτώχεια είναι ένα από τα θέματα τα οποία πιέζουν περισσότερο. Ε, επίσης, η αξιολόγηση για τι πολιτικέ θέσει Πέδρου θα πρέπει πιστεύω να εστιαστούν ει μια προσέγγιση επιτέλου του αποτελέσματο και να λάβουν υπόψη αυτό το, το, το, χαρακτήρα των στόχων και των μεθόδων τη μέτρησης και αποτίμηση επίση θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των κονδυλίων του προπολογισμού επί τη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και επίση να είναι οι δείκτε, οι μεταλλητές, κάτι όπω το ΑΕΠ κατά κεφαλή. Και επίση θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι πολιτικές θα ενταχθούν θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ομπρέλα κοινή, σε μια κοινή πολιτική. Και αυτό ε, συστήνοντας, συγκροτώντας ένα καινούργιο ταμείο. Τελευταίο, αλλά σημαντικό, εγώ θα σας τόνιζα ότι κάποιο μέλλον θα πρέπει να αναγνωρίσει την ποικιλία, την πολυμορφία της Γεωργίας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει επομένως να υπάρχει διαφοροποιημένη προσέγγιση και όχι ενιαία προσέγγιση για όλους και για όλα. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ στις διαβραβημένες παρουσιάσεις. Περιμένω να βάλω το ακουστικά γιατί μιλάω σουηδικά και δεν με καταλάβετε. Λέω ξανά ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες αυτές τις παρεμβάσεις. Καμιά φορά ήταν και αφιλεγόμενες μάλιστα. Πολύ χρήσιμο αυτό για μας. Που είναι τελευταία αναλύση, θα πρέπει να συναποφασίσουμε. Είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα κάτω από διαφορετικές ε, οπτικές γωνίες. Γιατί στο κάτω-κάτω η δημοκρατία είναι ε, μια προσπάθεια ισορροπίας και συμβεβασμό. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συγητή μας, τον κύριο Ντες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κύριοι εμπειρογνώμονες. Η ακρόαση σήμερα, όπως είπε και η πρόεδρος, μας προσέφερε πολλές νέες ιδέες και σκέψεις και ήταν πολύ πιο επικοδομητική από την περασμένη ε, ακρόαση. Είμαι κάπως αβεβαίως όσον αφορά κάποιες από τις δηλώσει. Ο κ. Λάγκμαν αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα σχετικά με τα δημόσια αγαθά και άλλοι το ανέφεραν αυτό και πού θα πρέπει να τοποθετήσουν αυτά τα δημόσια αγαθά. Στη δική μου έκθεση Έχω την εντύπωση ότι εν αντιθέσει προς την Κομισιόν θα πρέπει να τα βάλουμε στον πρώτο αλλά στο δεύτερο πυλώνα γιατί έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να ε, τα αξιολογήσουμε καλύτερα γιατί αν έχουμε ε, α, σφαιρική προσέγγιση για τους πυλώνες δεν θα μπορέσουμε παρά να τους ε, ε, λάβουμε υπόψη μας και σφαιρικά. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η αγροτική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωματική γραφειοκρατία για τους παραγωγούς, νέα συστήματα διαχείρισης, νέα συστήματα ελέγχου και άρα και νέους μηχανισμούς κυρώσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να ξαναρωτήσω τους συζητητές, ε, τους εμπειρογνώμονες, θέλετε μεταξύ του πρώτου πυλώνα που αναφέρονται γενικά οι, ε, τα, πληρωμές για τα, <clears throat> την προσφορά της Ευρω... Ευρωπαϊκής Γεωργίας να αποχωριστεί τελείως από το δεύτερο πυλώνα όπου θα μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την απόδοση κάθε παραγωγού αν κατάλαβα σωστά, τον καθηγητή Λάνεμαν, εάν υπάρχει μεταφορά χρημάτων από το πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να μπορεί να γίνει χωρίς συγχρηματοδότηση αυτό. Και θα ήθελα να ακούσω από τον τελευταίο εμπειρογνώμονα που αναφέρθηκε στην Ήπεθρο. Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο πρέπει να είναι ξεχωριστό το ταμείο εδώ ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να μείνει στην αγροτική πολιτική, αλλά εδώ οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε συγχρηματοδότηση. Δεν ξέρω από πού προέρχεται ο εμπειρογνώμονας αυτός, αλλά εγώ είμαι από μια περιοχή που επί 40 χρόνια ήταν πολύ καθυστερημένη στη Γερμανία και προχώρησε μόνο γιατί ακριβώς βελτιώθηκε η υποδομή εκεί. Δηλαδή, εάν έχουμε σήμερα στην Ευρώπη περιφέρειες με φτώχεια, όπου οι άνθρωποι υποφέρουν. Η δική μου εμπειρία είναι ότι θα πρέπει εκεί να επενδύσουμε στις υποδομές. Βέβαια θα μπορεί να υπάρχει και κάποιος συνδυασμό. Διαστρωτικά μέτρα και ύπεθρο. Διαστρωτικά μέτρα από ένα άλλο ταμείο βέβαια. Και θα είχα μετά και μια ερώτηση. Πώς φαντάζονται οι εμπειρογνώμονες αυτές στο μέλλον την απλούστευση του συστήματος. Εγώ θα ήθελα να ενταχθεί αυτή η απλούσευση στην έκθεσή μου. Έλαβα υπόψη ότι και είχα κάποια προβλήματα στην έκθεσή μου αυτό, ότι η ανακοίνωση λέω της Κομισιόν σε μεγάλους τομείς είναι πολύ ασαφής και δεν ενδείκνεται σαν βάση που θα βοηθήσει το Κοινοβούλιο να αναπτύξει το θέμα. Και θα ήθελα να το πω στους συναδέλφους. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε την απόφαση. Δεν επιτρέπεται να έχουμε ασαφή έκθεση που είναι ελεύθερη ε, που αφήνει την Κομισιόν απόλυτα ελεύθερα. Εγώ θα προσπαθήσω στην έκθεσή μου να έχω τις επόμενες μέρες περισσότερες λεπτομέρειες και που θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε έντονες συζητήσεις. Αλλά δεν θέλω να έχω μια έκθεση επιπόλαια που θα ασχολείται γενικά με την αγροτική, μελλοντική αγροτική πολιτική θα τύχει μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο γιατί δεν θα λέει πολλά πράγματα θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν και οι ευρωγνώμονε το βλέπουν τα πράγματα όπω εγώ, ότι εμεί ω κοινοβούλιο πρέπει να πούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε η Κομισιόν να έχει μια καλή βάση για την νομοθετική της έκθεση. Αυτά αρχικά. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Και τώρα ο Λουίς Καπούλα Σάντος. Muito obrigado, Presidente. Eu agradeço ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όχι μόνο για την παρέμβασή τους, τους ε, πυρογνώμονές μας, αλλά και για τα εκθέσει που μας έδωσαν, που θα μας χρησιμεύσουν ιδιαίτερα για τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με τον κύριο Ντες για την έκθεση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σημείο κύριο όσον αφορά αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι το νέο σύστημα των ενιαίων πληρωμών. Ο κύριος Στάγκερμαν μας παρουσίασε εδώ την εργασία του και εγώ θα ήθελα να δηλώσω τη διαφωνία μου και είναι δυνατόν να μου κάνει κάποιες αποσαφηνήσεις. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Στάγκερμαν είπε πως οι ενιαίες πληρωμές ε, εξυπηρετούν τη στήριξη των ε, εισοδημάτων και όχι την ανταμοιβή για δημόσια αγαθά και ότι θα ήταν υπέρ μιας ε, κοινή γεωργικής πολιτικής που θα βασίζεται μόνο στο δεύτερο πυλώνα και θα συγχρηματοδοτείται. Εγώ συμφωνώ με αυτό, γιατί η πρόταση της Κομισιόν να βάλει οικονομικά στοιχεία ε, όπως τα δημόσια αγαθά και να συμπληρώσει τα δημόσια αγαθά με περιβαλλοντικά θέματα κτλ. είναι υπέρ ε, Ε, της κοινοτική μεθόδου που ήδη έχει εκφραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Το νέο μοντέλο θα μπορούσε να αυξήσει την νομιμότητά του απέναντι στον ΠΟΕΜ αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό εγώ ήθελα να μου επιβεβαιώσει αυτή την προοπτική. Γιατί ούτως ή άλλως εγώ δεν βλέπω το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να γίνει ει βάθο συζήτηση ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ, Λουί, ο κύριο Χόφμαν. Και εγώ πιστεύω, όπω είπε και ο εισηγητή Αλβερτές, ότι σήμερα ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ε, παρουσιάσεις. Ίσως πιο ενδιαφέροντα από ότι έγινε με πριν μερικέ μέρε που είπαμε οι μέντσους αυτά που όλοι ξέραμε. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα βρήκα αυτά που είπε ο καθηγητής Τάγκαμαν και την του το ξεκαθαρό του συμπέρασμα ότι ας κάνουμε στη δεύτερη πυλώνα την πολιτική που αρμόζει στον δεύτερο πυλώνα. Γιατί να κάνουμε τώρα το πρασίνισμα αυτό στον πρώτο πυλώνα. Πιο λογικό θα ήταν να δούμε τι έχουμε στη σημερινή πολιτική στον δεύτερο πυλώνα και τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για την περιβαλλοντική πολιτική. Εσκύπτ κράτη-μέλη που περιέργω στο 95% των αγροτικών τους δαπανών τα δαπανούν στον πρώτο πυλώνα. Εκεί δεν υπάρχει δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας και γι' αυτό δεν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική ή προστασία στον δεύτερο πυλώνα. Θα ήταν λοιπόν καλό κάποια στιγμή να σκεφτούμε κατά πόσον το περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα για την γεωργία που υπάρχει σήμερα να το καταστήσουμε υποχρεωτικό και να το προωθήσουμε και εκεί που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό κάποια στιγμή. Να ενδυναμώσουμε δηλαδή το σημερινό μοντέλο, να το αναπτύξουμε. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή Τάγκαμαν. Να μην αναμειγνύουμε δηλαδή πράγματα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Το θέμα της απλούστευσης για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, πολύ καλά νομίζω το παρουσίασε ο καθηγητής Τάνγκαμαν. Δεν θέλουμε καταποκοπή ποτσά για τις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, αλλά να δούμε τι γίνεται με διοικητικά μέτρα. Θα μπορούσαμε να έχουμε παραδείγματος χάνει πολυετής πληρωμές, ε, ξέρω εγώ. Ίσως θα πρέπει την πληρωμή αυτή να την παίρνουμε μία φορά τα πέντε χρόνια. Να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αποτελεσματικά την γραφειοκρατία. Τέλος, όσον αφορά και τις τρεις τώρα παρουσιάσεις, ε, Χαιρετίζω ιδιαίτερα ότι αναφέρθηκε το θέμα της φτώχειας ε, στην αγροτική πολιτική. Αυτό που μου έλειψε όμως ήταν κάποια αναφορά όσον αφορά την γύρανση στις αγροτικές περιοχές. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που ούτε και η Κομισιό το ανέφερε και ούτε και εμείς φαίνεται το αναφέρουμε πάρα πολύ, αλλά που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Σικερέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τόσα πολλά πρέπει να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε μετά από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Εγώ διάβασα όλα τα οποία μέσα σπίγει ο ε, θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε όμως παρόλα αυτά είναι αλήθεια ότι, ότι υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες προκλήσεις και κάποιες που είναι όμως όχι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Ε, και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς για όλες αυτές τις δαπάνες θα υπάρξει η νομιμότης η κατάλληλη. Και αυτό και προτείνω να κάνουμε. Αυτό θέλω να κάνουμε. Δεν θέλω να επικρινώ κανέναν γιατί γνωρίζω και έχουμε τώρα μια πολιτική συγκυρία ιδιότυπη στην οποία δούμε και επομένως θα πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε και τόσα πολλά να αλλάξουμε γιατί οι τιμές αυτές είναι σταθερότητα για τους γεωργούς. Άρα θα πρέπει το επίπεδο των τιμών, το ιστορικό επίπεδο θα πρέπει να παραμείνει. ιστορική προοπτική μας οδηγεί σε μια τέτοια στάση. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο, όμως εισοδημάτων επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε τον προπολογισμό. Θα πρέπει ο προπολογισμό μα να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσουμε να επιτυχούμε του στόχου μα. Επίση, υπάρχει και ένα άλλο προβληματάκι. Το ότι έχουμε τόσου πολλού στόχου Όσον αφορά την ε, η ανάπτυξη της υπαίθρου, την κοινωνική πολιτική, την αλλαγή του κλίματο κλπ. Το οποίο όμω εκνευρίζει, το οποίο προβληματίζει του ε, φορολογούμενου. Δηλαδή έχουμε ε, ίσως μερική επικάλυψη των στόχων, το οποίο δεν είναι σωστό μια που το έχουμε τεθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρος κ. Σικέρσκη. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καλινόσκη. Σα ευχαριστώ. Ακούσαμε όλου αυτού του επιρρογνώμονε και είχαμε μέσα αυτή τη συγκεκριμένη την προσέγγιση του κ. Τάγκερμαν, ο οποίος, ο οποίος ενατένισε το μέλλον της γεωργίας μας και μας παρουσίασε το πώς εκείνος αξιολογεί τα πράγματα σε σχέση με το κείμενο της Επιτροπής. Νομίζω επομένως ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γεωργία μας γίνεται όλο ένα και λιγότερο ανταγωνιστική. Χάνουμε έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Επομένως, το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια Κατά πόσον που να βρούμε μια λύση, έστω και συμβαστική, κατά πόσο θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τη γεωργία μα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε εάν θέλουμε να είμαστε φιλικοί στο περιβάλλον, αν θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη κοινωνική πολιτική, εάν ή αν από την άλλη μεριά θέλουμε να παραιτηθούμε από αυτή μας την προσπάθεια και από ένα τέτοιο συμβασμό και γιατί αλλιώς θα βγούμε χαμένοι για την επόμενη έπτα ετία. Οπότε τώρα όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές θα πρέπει να εξεταστεί τι θα γίνει σε σχέση με τα παλιά ή τα νέα κρατημέλη κατά πόσο δηλαδή θα έχουμε ισότητα καταβολής πληρωμών ή δίκαιες πληρωμές γιατί έχουμε βόρειους, νότιους, ορεινούς, παιδινούς έχουμε μέρη με καλό καιρό, με σκληρό καιρό και έχουμε και αυτή την έκθεση την οποία επιψηφίσαμε ή στο Κοινοβούλιο εκεί όπου μιλούμε για τα αντικειμενικά κριτήρια όμως σιγά σιγά αρχίζουμε και τα αγνοούμε. Θα πρέπει να τα θυμηθούμε αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια. Ο καθηγητής Στάνκεβαν επίσης μας ανέφερε την έννοια του ενεργού αγρότου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την έννοια και θα πρέπει να προβληματιστούμε διότι θα αφορά αυτό κάποιον ο οποίος κατέχει ένα κομμάτι γης και το καλλιεργεί. Βεβαίως μπορεί να το εκμισθώσει, όμως, εάν το εκμισθώσει μετά, θα αποκερδάνει το μίστομα για αυτή τη γη. Οπότε αυτό είναι πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλο είναι. Στην Πολωνία. Άρα, θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η κατανομή μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα όσον αφορά και τα κονδύλια και τα εργαλεία πολιτική. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεταξύ νέων παλιών κρατών μελών μεγάλη διαφορά αυτό το 20%. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ και τώρα να αποφασιστεί. Θα πρέπει να βλεπουμε πρώτα πρώτα υπόψη την ποικιλία του, το διαφορετικό χαρακτήρα της γεωργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις μικρές παρατηρήσεις να κάνω. Τα προβλήματα της συγχρηματοδότησης αναφέρθηκαν. Δεν ξέρω κατά πόσον οι εμπειρογνώμονε ε, έχουν κάποιες προτάσεις πώ θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συγχρηματοδότηση διαφορετικά για να ενδυναμώσουμε την ύπεθρο. Ότι κάτι πρέπει να γίνει είναι γνωστό. Γιατί, Γιατί η συγχρηματοδότηση θα είναι ένα κριτήριο αποκλεισμού. Δεύτερον, νομίζω ότι η παραγωγή είναι πολύ πιο ικανή να προσαρμοστούν στις ε, κλιματικές αλλαγές παρά να προσαρμοστεί η ύπεθρος στις ε, δημογραφικές αλλαγές. Γιατί ο ρυθμός των δημογραφικών αλλαγών είναι πάρα πολύ έντονος, ιδίως στην ύπεθρο. Πολύ πιο έντονος. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικός ο δεύτερος πυλώνας. Είναι το μέσο το ώστε πραγματικά να μπορέσουμε εκεί να δράσουμε ενισχύοντας γιατί τι ωφελεί στους παραγωγούς είναι μια ύπαθρο στην οποία είναι μόνοι τους. Και θα ήθελα να προσέξουμε με όλους τους στόχους που έχουμε μετά τα προγράμματα που θέλουμε να προωθήσουμε να μην ξεκινήσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί αν πολλά προσπαθήσουμε να κάνουμε δεν θα μπορέσουμε πια να ενισχύσουμε. Να μην είμαστε δηλαδή πολύ ευραίος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Άγνιο, γρήγορα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας. Πολλά σχόλια έγιναν αποκλειστικά για την δεύτερο πυλώνα που νομίζω ε, μπορώ να δώσω 50-60 παραδείγματα, θα σας δώσω μόνο τρία. Προώθηση των της ελληνικής πατάτας στη Σουηδία. Η Σουηδία έχει τη δική της πατάτα, δεν το χρειάζεται αυτό. Έχει γίνει φοβερή κατάχρηση του δεύτερου πυλώνα χρήματα στι ισπανικέ επιχειρήσει που ούτε καν υπάρχουν, κατασπατάληση χρημάτων. Την περασμένη φορά στην Ολομέλεια στι Βρυξέλλε ανέφερα τους Ούγκρους, τους Ουγγρικούς σκύλους όπου δήθεν δίνονται ένα σωρό λεφτά για να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων, δίνονται τα χρήματα, αλλά η ζωή παραμένει σκυλίσια για τους ουγγρους σκύλους. Απασχόληση. Περισσότερες χώρες έχουν το εσύ δηλαδή την, ε, το φόρο απασχόληση, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να πληρωθούν οι δουλειέ στην ε, Ήπεθρο. Μετά, για τους αποτεφρωτές, γιατί να μην επιχορηγηθούν και αυτοί. Και έπειτα, η νέος κανονισμός για την Ένωση για την αποθήκευση των, του χείριου κρέατος, του βόηου κρέατος, ε, να χρηματοδοτηθούν και αυτά. Και τώρα, υγεία και ασφάλεια οι γερικές εκμεταλλεύσεις, ε, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, ε, ειδικά ε, κράνη πρέπει να προβλεφθούν και προστασία για τους εργαζόμενους στις εκμεταλλεύσεις. Ο Μάρτιν Όσλινγκ. Σύντομα. Κύριε είπατε ότι αν έχουμε ε, την αλλαγή του επαγγέλματο στο στον πρώτο πυλώνα, δεν θα είναι αυτό συμβατό με τον ΠΟΕ. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Επίσης, λέγεται ότι θα πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμέ σύμφωνα με την μονάδα δημοσίου αγαθού. Τι σημαίνει αυτό, πώς θα το μπορέσω να το ε, να το ορίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, εάν δεν έχουμε πράσινη, πράσινο πρώτο πυλώνα και προσπαθήσουμε να διορθώσουμε με το δεύτερο πυλώνα ότι δεν έχει πάει καλά, δεν μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει να φροντίσουμε καταρχήν να έχουμε μια αγροτική πολιτική η οποία να είναι σύμφωνη με αηφόρο γεωργία. Και στους δύο τομείς. Και όχι μόνο για διευθυντές. Ευχαριστώ. Μάρτιν. Καλνιάτη και μετά Νίκολσον. kungs. Ε, es gribēju par ε, tiešajiem maksājumiem, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις άμεσες πληρωμές. Για ε, την Γεωργία στην Λετωνία είναι το πιο σημαντικό σημείο αναφέρθηκε αυτό ότι θα πρέπει να αποτελέσει, μάλλον το τι θα είναι η, βάση για τις πληρωμές αυτές στην ε, Λετωνία για πάρα πολλές, χώρες, για πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις. Η κοινή χειρική πολιτική δεν θα ήταν τίποτα χωρίς αυτές τις άμεσες ε, πληρωμές. Θα πρέπει να υπάρχει γενικά ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ένωση. για την ώρα προτείνουμε ε, εμεί σε περισσότερη σαφήνεια στο σύστημα, γιατί η ενιαία πληρωμή θα είναι χαμηλότερη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτό κάπως να το αντισταθμίσουν. Αν μιλάμε για το 75% της μέσης πληρωμής, Εμείς ε, θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι το μάξιμο με 120% για να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας. Φυσικά και χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια. Και το ανέφερε και ο κύριος ε, Γιάμπορ, ότι πρέπει κανείς να δει τον πληθυσμό, τη διαθέσιμη γη στις περιοχές της Υπέθρου, Εάν θέλει κανείς δηλαδή να διατηρήσει την γεωργική γη, θα πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής. Θα πρέπει να βελτιωθεί το, το ανθρώπινο υλικό και οι τεχνικές δυνατότητε. Ευχαριστώ. Τζιμ Stinkerson. The, the division between the first pillar and the second pillar, and this is where the battleground εδώ έχει γίνει πολλή ε, λόγος για το δεύτερο πυλώνα και πιθανότατα πολλά πράγματα δεν θα είναι στη μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι η μετακίνηση, ας πούμε, να να μιλήσουμε για νέα πληρωμή. Παλιά υπήρχε μια πληρωμή για το ε, μικρό, μια πληρωμή για κάθε ζώο, μια πληρωμή για κάθε δέντρο κτλ. Και μετά πήγαμε στην ενιαία πληρωμή. Να το συνεχίσουμε αυτό ή να βάλουμε μια άλλη αναφορά. Όλοι δέχονται ότι δεν μπορεί κανείς να πληρώνεται ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε μία περίοδο αναφοράς. Ίσως αυτός ήταν καλύτερος τρόπος για κατανομή των κονδυλίων. Και έπειτα να ρωτήσω, αυτό που είδα εγώ, πείτε μου αν κάνω λάθος, η βιομηχανία βοήου και γιου κρέατος ε, ε, είναι σε, ε, σε ύφεση από τότε που εισήχθη η ενιαία πληρωμή. Έχω δίκιο ή όχι. Φταίει αυτό. Και έπειτα, πολιτική για γεωργία. Δεν είναι η περιβαλλοντική πολιτική, ούτε η κοινωνική πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντο, το τελευταία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τι πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Θα ήθελα να στραφώ προ τον καθηγητή Τάνεμαν. Κύριε καθηγητά, στην ε, παρουσίασή σα είπατε ότι έχετε αμφιβολίε για τι άμεσε πληρωμέ. Είπατε ότι δεν σχετίζονται άμεσα με την ε, τροχική ασφάλεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί σε ορισμό τομεί έχουμε μια ε, εγκατάλειψη ε, συνεχή, δεν θα ήταν καλό να υπήρχε μια άμεση πληρωμή για να διατηρηθεί αυτή η παραγωγή. Επίση είπατε ότι οι άμεσε πληρωμές σχετίζονται και με τι ψηλέ τιμέ. Εγώ ξέρω όμω, ότι τουλάχιστον στη Γερμανία 11% μόνο του εισοδήματο ε, δαπανούνται για τρόφιμα. Αυτό δεν μου φαίνεται υπερβολικά υψηλό, των αντίον. Νομίζω θα ήταν καλό να περάσουμε σε πιο υψηλά επίπεδα, να δαπανούμε δηλαδή περισσότερα χρήματα για καλά τρόφιμα. Το σημαντικό μου ερώτημα είναι το εξή. Πολύ καλό που είπατε ότι ε, είναι καλό να είμαστε δίκαιοι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, δικαιοσύνη όσον αφορά τα εισοδήματα. Αυτό πώς το εξηγείτε. Δηλαδή να συγκρίνεται με την κοινωνική ασφάλεια ο κάθε παραγωγό να περιγράφει ποια είναι η κατάσταση του εισόδηματό του, δηλαδή πώς θέλετε να το επιβάλλετε αυτό. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να ζητήσουμε να συγχωρήσουν οι διερμηνείς ε, γιατί ακόμα ένα λεπτάκι θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει να είστε οι υπόλοιποι που έχετε το λόγο να απαντήσετε οι τρει προσκεκλημένοι μα Πάρα πολύ δεν έχουμε χρόνο πρώτα πρώτα κύριο Στάνγκεμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ιδέες. Λόγω του περιορισμένου του χρόνου δεν μπορώ πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτά. Το βασικό θέμα πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τα δημόσια αγαθά στον πρώτο ή στο δεύτερο πυλώνα, για μένα είναι ξεκάθαρο. Δεύτερος πυλώνας γιατί μόνο στο δεύτερο πυλώνα μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τόσο όσο χρειάζεται για την προσφορά δημοσίων αγαθών. Γιατί κάθε εκτάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν συμβάλλει κατά τον ίδιο τρόπο στο δημόσιο αγαθό. Και γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε. Γι' αυτό λέω δεύτερος πυλώνας. Κατά με λοιπόν μια πολιτική η οποία θα κινώ, το περισσότερο προς μια εστίαση που μετέφερε μετά από τον πρώτο πυλώνα προς τον δεύτερο πυλώνα καλύτερη. Αμέσως τίθεται λοιπόν το θέμα της συγχρηματοδότησης. Εάν κάνουμε αυτό που είχαμε στην πολλαπλή συμμόρφωση στο παρελθόν, δηλαδή ένα ευρώ από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα και μετά συμπληρωματικά τα εθνικά κονδύλια, αυξάνεται το όγκος τεράστιο. Δεν θα πρέπει ο στόχο μας να είναι να δαπανίσουμε ακόμη περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει ένα άλλο σύστημα. Καταρχήν, και θα με η επαναστάτη που θα σα τα πω αυτά, είναι σωστό τα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτούν γιατί θα θέλουν και να συναποφασίζουν πού χρειάζονται πια δημόσια αγαθά. Και για να μην είναι προστατικά τα ποσά αυτά, θα ήταν καλύτερο οι οικονομικές συμβολές ε, των κρατών μελών στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθούν και τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για μια συγχρηματοδότηση στο δεύτερο πυλώνο. Και έτσι θα υπάρχει και συν υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων για το δεύτερο πυλώνο. Ε, τι σημαίνει η μονάδα του δημοσίου σύμφωνα με την θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρήματα. Βέβαια αυτό είναι ένα ένας πολύ σύντομος ορισμός από μένα, αλλά ακριβώ αυτό γίνεται στο δεύτερο πυλώνα και το αποτελεσματικό είναι ότι θα πρέπει σημαντικά να δεσμευτούν τα κονδύλια αυτά. Θα υπάρχει δηλαδή μια σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και του δημοσίου που θα ορίζει τι θα πρέπει να προσφέρει ο παραγωγός ο οποίο θα πληρώνεται για τη συγκεκριμένη αυτή συμβολή του. Δεν θα μπορεί να υπολογιστεί αυτό ανατόνο ίσως, αλλά θα είναι σημαντικό να οριστεί η απόδοση και θα υπάρχει μια σύμβαση που θα υποχρεώνει τον παραγωγό ακριβώς αυτό να το προσφέρει που έχει υπογράψει εκεί. Θα πρέπει να συζητήσουμε ίσω ε, πώ θα ορίσουμε το ύψο των πληρωμών αυτό. Δεν θέλω να επιστρέψω στι λεπτομέρειε. Υπάρχουν διάφορε διαδικασίε με τι οποίε γίνεται κάτι τέτοιο θαυμάσια. Μετά ερωτήθη γιατί η αλλαγή της καλλιέργειας δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό δεν είναι θέμα συμβατότητας με τον ΠΟΕ, αλλά οι άμεσες πληρωμές αυτή τη στιγμή κοινοποιούνται στον ΠΟΕ ότι πέφτουν δηλαδή στο πράσινο κουτάκι και αν οι άμεσε πληρωμέ αυτέ θέλουμε να μπουν στο πράσινο αυτό κουτάκι, δεν επιτρέπεται να είμαστε προκλητικοί. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει ο παραγωγός να παράγει για να πάρει τι πληρωμές αυτές. Γιατί αλλαγή, αλλαγή της ε, καλλιέργειας δεν, ε, ε αλλαγή της σημαίνει άμεσα παραγωγή. Γι' αυτό μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με το πράσινο κουτάκι της, ε, του ΠΟΕ. Μετά ερωτήθη και τελειώνω εδώ πρόεδρε. Ρωτήθηκε κατά πόσον δεν είναι σημαντική η ε, αποχώρηση από την Ήπεθρο ένα πρόβλημα για την παραγωγή τροφίμων. Αυτό όμως ε, δεν είναι ένα πρόβλημα γιατί δεν φεύγουν οι, οι εκτάσεις οι καλλιεργούμενες. Αυτή η με η μετανάστευση δεν έχει επίδραση πάνω στην αγροτική παραγωγή. Τα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι εμείς θέλουμε στο μέλλον να κατανοίγουμε τις άμεσες πληρωμές δίκαια. Μα αυτό θα είναι θέμα πραγματικά ε, δικαιοσύνης. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το εισόδημα του ε, παραγωγού. Φαντάζομαι ότι η Βασίλισσα της Αγγλίας δεν χρειάζεται άμεσες πληρωμές, αλλά φτωχοί παραγωγοί το χρειάζονται. Δεν μιλάμε εδώ για με, ε, για άτομα και για εισοδήματα. Βίνσεντ, σε παρακαλώ, εσύ έχεις το λόγο. Ναι, 45 δευτερόλεπτα θα μιλήσω μόνο. Καταρχήν πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Και πίσω από τις μεγάλες ιδέες αυτό που είναι σημαντικό είναι αν επιθυμούμε νέου να ανακατανύμουμε τα, την ε, διάταξη για να την προσαρμόσουμε στην πτυτικότητα των τιμών. Και έπειτα, η δεύτερη ιδέα, είμαι υπέρ, βέβαια διαφωνώ ίσως, αλλά είμαι υπέρ του να υπάρξει στον πρώτο πυλώνα ένα είδος πρασινίσματος. Ακόμα και αν είναι διαφορετική η μεταχείρισή του με, από τα μέτρα για την ανάπτυξη του ισηπέθρου πάντως ε, ο έλεγχος υγείας της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής μας έδωσε κάποια κριτήρια που επιτρέπουν να δώσουμε περισσότερο νόημα στον πρώτο πυλώνα. Και έπειτα πιστεύω πως θα πρέπει να είσαστε να υπαγρυπνείτε όσον αφορά την θέσπιση ανώτατων ορίων καθώς και στον ορισμό του ποιο χέρι της δημόσιας στήριξης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε Βίντσεν. Και τώρα τελευταίος ο κύριος Τζαμπόρα. Uh, ε, έχω κάποιες παρατηρήσεις να αφορά τη σχέση μεταξύ της πολιτικής ανάπτυξης και της γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι πολιτικές αυτές δεν θα πρέπει μόνο να αφορούν τη γεωργία. Η γεωργία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών, αλλά νομίζω ότι πέραν αυτές τις πολιτικές υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα το, της υπαίθρου έτσι. Γι' αυτό σας λέω, θεωρώ ότι αυτές οι πολιτικές που να λάβουν υπόψη όχι μόνο τη Γεωργία, που είναι όμως αναπόσπαστο σημαντικό τμήμα τους. Τώρα, όσον αφορά την απλούστευση της μεθόδου αξιολόγησης, θεωρώ ότι για να απαντήσω και σύντομα αυτό που πρώτο που θα πρέπει να προσθέσουμε τους δείκτες. Πάνω από 100 είναι. Να το απλουστεύσουν. Και αυτό είναι σημαντικό. Το σύστημα αξιολόγησης δεν αποδίδει κάρπου σήμερα. Δεν λειτουργεί σωστά. Πολλές φορές απλώς τσεκάρουμε διάφορα <clears throat> έντυπα γύρανση του πληθυσμού της υπαίθρου, όπως είπατε σωστά, υπάρχει σχέση για την αύξηση του υπαίθρου και του δημογραφικού εκεί πέρα. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και αυτό το η Ένωση, Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλους ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονές μας, αλλά και για την η έντονη συζήτηση που έγινε μας δείχνει ότι σίγουρα πρέπει πολλά να σκεφτούμε μου έρχεται να πω με ένα σύντομο σχόλιο στα τελευταία που είπε ο κύριο Τάγκερμαν, ο καθηγητής Τάγκερμαν. Ίσως το Αμερικανικό Κογκρέσο ποιος ξέρει πώς θα είχε αντιδράσει στην παρέμβαση του κύριου Τάγκερμαν. Η Επιτροπή Γεωργίας του Κογκρέσου θα είχε ίσως αντιδράσει διαφορετικά από το πώς αντιδράσαμε. Εμείς ευχαριστούμε τους υπηρεγνώμενους, τους καθηγητές και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίαση που προβλέπεται για τι 28 Φεβρουαρίου στι 3 τέλο συνεδρίασης. Μας συγχωρείτε